Uh, dear κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται στους φακέλους σας. Θέλετε να αλλάξουμε κάτι, δεν βλέπω κάποια πρόταση. Αναγγελής Πρόεδρου. Τρεις. Η συνεδρίαση τη Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την προστασία στο διαδίκτυο του ιδιωτικού βίου με την ενίσχυση των συστημάτων ηλεκτρονικής και την αυτονομία των συστημάτων ηλεκτρονικής τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συμμετέχει και η Επιτροπή μα, θα διοργανωθεί στι Βρυξέλλες στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2015. Ενδιαφερόμενοι βουλευτέ τη Επιτροπής μας ε, είναι θερμά ευπρόσδεκτοι. Ε, θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη διάσκεψη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την προστασία του ιδιωτικού βίου στο διαδίκτυο. Δεύτερο σημείο, ο Επίτροπος Μοέδας θα είναι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών, ελέγχου των προπολογισμών, Κοκοβού, την 5η, 3 Δεκεμβρίου, από τις 3 στην αίθουσα 5G3 στο κτίριο Αρτιέρο Σπινέλη για ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την απαλλαγή του 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο, ο Επίτροπος Μοέδας ε, ασχολείται και με δικά μας θέματα εντός του παιδιού των αρμοδιοτήτων μας, όπως η, Επιτροπή, η πολιτική κοινοτομία και το καθεξής. Τρίτο σημείο, η συνεδρίαση της Επιτροπής μας την 3η-1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί διότι θα προηγηθεί θα προηγηθεί από τις 9 στις 10 συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Αυτά είναι τα νέα. Εάν έχετε κάτι επιπλέον, κάποια αναγγελία, κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Ντανίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω την ε, στήριξή σας και κάτι κατεπήγον που θα ήθελα να προσθέσουμε στην μέση διατάξη. Την ερώτηση που απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μένα και τον κύριο Κάριν υπογεγραμμένη στις 21 Οκτωβρίου φέτος, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε ακόμη απάντηση για το σύστημα ανταλλαγής εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Θα ήθελα λοιπόν, αν γίνεται, να συμπεριλάβουμε στη μέση διάταξη αυτή την ερώτηση για το ETS. Είναι ερώτηση από μένα και τον κύριο Κάριν, που αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μα. Δυστυχώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η προθεσμία για να δοθεί απάντηση από τη σκοπιά των δικών μας κανόνων τουλάχιστον ήταν 16 Νοεμβρίου, πριν από 10 μέρες δηλαδή. Ωστόσο, δυστυχώς. Η προθεσμία αυτή δεν είναι υποχρεωτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Επίτροπος Καλνιέται. ενημέρωσε ότι η απάντηση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και θα αποσταλεί στο Ευρωκοινοβούλιο ε, συντόμως. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν δεν λάβουμε απάντηση στα τέλη αυτής της εβδομάδας ή στην αρχή της επόμενης, τότε ας αποφασίσουμε ότι το θέμα αυτό θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη αλλά τη επόμενη ε, συνεδρίαση τη Επιτροπή Ήτρε. Η στην αρχη της επομενης τοτε ας αποφασισουμε οτι το θεμα αυτο θα περιληφθει στην ημερησια διαταξη της επομενης επομενη της επιτροπης επιτροπη ητρε η αντιδραση μας σε μια τέτοια κατάσταση είναι να συμπεριλάβουμε ένα συγκεκριμένο σημείο για να συζητηθεί το θέμα ETS πριν τα Χριστούγεννα. Ε, στη συνεδρίαση πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι έχουμε κι άλλη μία. Έχουμε μια κοινή συνεδρίαση πριν τα Χριστούγεννα νομίζω. Θα σκεφτούμε λοιπόν αν ε, θα χρειαστεί να το συμπεριλάβουμε. Και ε, αυτή τη στιγμή το έχει σημειώσει η γραμματεία της Επιτροπής μας για τις επόμενες ημερομηνίες συνεδρίασης. Ο Επίτροπος Καλνιέται όμως είπε ε, συντόμως Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το σχολείο σας. Κάποια άλλη παρατήρηση, συνάδελφοι. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, σχόλια, οπότε να πάμε στο τέταρτο σημείο. Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τροφοδοσίας των Σιδηροδρόμων. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Η ανταλλαγή αυτή απόψεων με τους εμπειρογνώμονέ μας που είναι απέναντί σα συνάδελφοι, είναι απλώ η αφετηρία της εργασία της Επιτροπής μας για την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρόμων. Να καλωσορίσω τους ομιλητέ μας και σα ευχαριστώ και τους δύο για την προθυμία σας να παραβρεθείτε. να αναγγείλω ότι κάθε ο μιλητής θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση και καλό θα ήταν να μπορείτε να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. Παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς έχετε και το χρονόμετρο στην οθόνη, οπότε μπορείτε να κοιτάτε κι εσείς το χρόνο και να είστε βέβαιοι ότι όλα πάνε καλά. Θα Έχουμε συζήτηση αμέσως μετά τις ε, εισηγήσεις σας. Να ξεκινήσω, να ξεκινήσω με τον κύριο Φιλίπ Σιτροέν. Είστε Γάλλος? Σιτροέν. Μάλιστα. Γενικός Διευθυντής της UNIFE Εάν θέλετε ε, να μας συστηθείτε εσείς ο ίδιος, διότι δεν έχω μπροστά μου το βιογραφικό σας σημείωμα, οπότε ε, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Μπορεί να εργαστήκατε για την ίδια την ε, Citroën. Λόγω του ονόματος ε, μπορεί να έχετε κάποιες σχέσεις με την εταιρεία αυτή. Λίγα λόγια για τον εαυτό σας παρακαλώ, λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, θα απαντήσω σύντομα. Είμαι γονός του ιδρυτή των εργοστασίων Citroën, αλλά έρχομαι εδώ εκ μέρους της σιδηροδρομικής βιομηχανίας. Δεν ελέγχει εξάλλου η οικογένεια Citroën εδώ και δεκάδες χρόνια την αυτοκινητοβιομηχανία Citroën. Δουλεύω λοιπόν στους σιδηρόδρομους. Για χρόνια ήμουν σύμβουλος εδώ όσον αφορά του σιδηρόδρομους στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Ε, δούλεψα και με τον άλλο Υπουργό Μεταφορών. Για χρόνια ήμουνα στην ΕΡΑΤΕΠΕ, είναι το αντίστοιχο της ε, ΣΤΙΠ, στο Παρίσι, δηλαδή πρόκειται για τις ε, μεταφορές στην πόλη του Παρισιού. Μετά δούλεψα και στην SNCF, τα τρένα δηλαδή τα γαλλικά. Και μετά έκανα μια εταιρεία που ονομάζεται Στράκ, είναι πολύ γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τους σιδηρόδρομους και στη συνέχεια ε, δούλεψα με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές ε, για εξοπλισμό σιδηροδρόμων. Αυτά έκανα τα τελευταία 30 χρόνια λοιπόν. Πρόεδρε, θα πω δύο λόγια στα γαλλικά, ευχαριστίες βασικά για να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας κάλεσε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ επίσης και την Ευρωβουλευτή Μαρτίνα Βέρνερ και όλους τους Ευρωβουλευτές εδώ παρόντες. Όλους ιδιαίτερος όμως ευχαριστώ την Μαρτίνα Βέρνερ η οποία ε, δουλεύει πάνω στην έκθεση αυτή για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συνεχίσω μετά από αυτά που σας είπα πριν για το τι είναι η, ο κλάδος των σιδηροδρόμων και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Σήμερα μου δίνεται ευκαιρία να σας πω περισσότερα για τον κλάδο μας και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας στην Ευρώπη και γενικότερα. Το ερώτημα, λοιπόν είναι τι ακριβώς είναι ο ευρωπαϊκός κλάδος προμήθειας σιδηροδρομικού εξοπλισμού όπως γνωρίζετε, πρόκειται για τους πελάτες από τη μια μεριά, τη διαχείριση των υποδομών και από την άλλη μεριά έχουμε τον εξοπλισμό σιδηροδρόμων. Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που οφείλεται στις πολυάριθμες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Τα βλέπετε και στην ε, διαφάνεια. Έχουμε είτε το τροχαίο υλικό, είτε την ε, σήμανση και σηματοδότηση και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και τον ρόλο που παίζουν οι διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ε, τομέα, είτε πρόκειται για τα τρένα υψηλής ταχύτητας, είτε πρόκειται για άλλες αγορές στην πόλη. Υπάρχουν επίσης πολλά μεγέθη επιχειρήσεων. Όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου γίνεται η συναρμολόγηση από κοινού, έτσι και στους σιδηροδρόμους έχουμε διάφορα συστήματα συναρμολόγησης, δηλαδή χρησιμοποιούμε υλικό από διάφορες πλευρές και το συναρμολογούμε. Είναι αυτό που ονομάζουμε System Integrators. Είμαστε ένας πανευρωπαϊκός κλάδος Γαλλία, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Τσεχία είναι χώρες που έχουν μια μεγάλη βάση και παράδοση ε, βιομηχανίας όσον αφορά τον εξοπλισμό σιδηροδρόμων. Τώρα, γιατί είναι στρατηγική σημασία ο κλάδο αυτός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αρχίζουν επίσημα σήμερα στο Παρίσι διαπραγματεύσει για το COP21. Επιτρέψτε μου να σα θυμίσω ότι συνεισφέρουμε και εμείς την ανάπτυξη ενός πιο φιλικού για το περιβάλλον τρόπου μεταφοράς, σιδηρόδρομη δηλαδή, γιατί όμως είμαστε ένας εμβληματικός για την Ευρώπη κλάδος. Πρώτα απ' όλα είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη. Πάνω από 400.000 άνθρωποι απασχολούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη στον κλάδο αυτό. Δεύτερον, είμαστε ένας καινοτόμος κλάδος. Η καινοτομία είναι στο DNA του ευρωπαϊκού κλάδου και επενδύουμε σήμερα ένα μεγάλο μέρος του τζίρου στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έτσι προχωρούμε σε καινοτομία και έτσι και προχωρήσαμε στο τρένο υψηλής ταχύτητας, στο, στην ευρωπαϊκή διαχείριση σειροδρομικής κυκλοφορίας και διάφορα αυτόματα συστήματα, μετρό κλπ. Επίτα, είμαστε υπεύθυνη για την ε, ανάπτυξη όλων των συστημάτων σιδηροδρόμων. 47 δισεκατομμύρια ευρώ ο ευρωπαϊκός αυτός ο κλάδος σήμερα είναι υπεύθυνο για το 46% της αγοράς. Επίσης, η σημερινή συνάντηση μας δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε και για τις ευκαιρίες αλλά και για τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Τα καλά νέα είναι ότι η αγορά σιδηροδρόμων θα συνεχίσει να αυξάνεται σε όλες τις υπήρους. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία για απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό παγκοσμίω. Επειδή υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τάσεις της αστικοποίησης, αστιφιλίας, επειδή ε, υπάρχουν προβλήματα με την ενεργειακή προμήθεια και υπάρχει και ανησυχία για το περιβάλλον. Γι' αυτό θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του κλάδου 2,7% ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρά βέβαια τις οικονομικές αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκοσμίω. Φυσικά ε, υπάρχουν ε, και αλλού αντίστοιχε τάσει στην Βόρεια Αμερική, την Νότια Αμερική, η Ασία, Ειρηνικός και σε άλλες περιοχές του κόσμου που σημαίνει ότι είμαστε αντιμέτωποι και με ανταγωνιστές παγκοσμίω. Τώρα η πρόκληση ποια είναι. Επίτροπος Μπιενκόφσκα όταν είχε την ακρόασή της τον Οκτώβριο που μας πέρασε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να έχει πρόσβαση στις αγορές τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω. Αυτό είναι περισσότερο αληθές από οπουδήποτε αλλού στη δικιά μας την περίπτωση, στο δικό μας τον κλάδο. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι αγορές τις οποίες είχαμε άνετα πρόσβαση τα προηγούμενα χρόνια τώρα περιορίζονται περισσότερο και δεν είναι πια τόσο ανοιχτές ε, στον ευρωπαϊκό κλάδο προμήθειας όπως ήταν παλιότερα. Σήμερα μόνο 67% της συνολικής ε, αγοράς είναι το κομμάτι στο οποίο έχουμε εμείς πρόσβαση. Και η μείωση αυτή έχει να κάνει με άλλες αγορές όπως είναι η Κινέζικη, η Ιαπωνέζικη και εκείνη της Κορέας. Πολλές χώρες σήμερα εφαρμόζουν προστατευτικά μέτρα για να προωθήσουν και να προστατεύσουν τον χώριο κλάδο τους. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λοιπόν δεν έχουν πάντα ίση πρόσβαση σε διαγωνισμούς για προμήθειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, είναι ζωτική σημασία στις διαπραγματεύσεις που έχουμε τώρα για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ιαπωνία. Επίσης, ο κινέζικος παράγοντας, η δικιά τους αγορά που γίνεται όλο και πιο προστατευτική, οι άλλες αγορές όπως η Νότια Αφρική και η Ινδία απαιτούν τα εργοστάσια μας να εγκατασταθούν στις δικές τους τις χώρες για να προμηθεύουν τη δικιά τους αγορά. Ας δούμε λιγάκι τώρα την πρόκληση που έχουμε και την απειλή από την ε, Ασία. Αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό από την Ασία, κυρίως από την Κίνα και την Ιαπωνία και μάλιστα όλο και περισσότερο. Αυτό φάνηκε και από την μελέτη επισκόπηση για το 2013 και τώρα δύο χρόνια αργότερα η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό από την Κίνα, Πολλοί από εσά έχετε ακούσει τα νέα πριν από λίγες εβδομάδες για τη συγχώνευση των δύο μεγάλων κατασκευαστών, της CNR Corporation και την CSR Corporation, που μαζί είναι 31 δισεκατομμύρια σε πωλήσει στις ΗΠΑ το 2013. Τώρα λοιπόν έχει φτιαχτεί μια νέα εταιρεία που είναι ε, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ε, τρένων στον κόσμο, η CRRC Corporation. Και ενώ λοιπόν ε, η κινέζικη, ο κινέζικος κλάδος είχε επικεντρωθεί στην κινέζικη αγορά, τώρα είναι παρόν και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική και στην Τουρκία και τώρα και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και ο επόμενος στόχος τους είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Μπορούμε να σας δώσουμε το παράδειγμα των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του 16 1 για μια νέα γραμμή ανάμεσα στη Βουδαπέστη και το Βελιγράδι, που από ό,τι φαίνεται θα φτιαχτεί από τους Κινέζους. Και τέλος εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι περισσότερα από τα συμβόλαια που παίρνουν τελικά οι Κινέζοι προμηθευτές συμπεριλαμβάνουν και επενδυτικά προγράμματα με κρατικές επιδοτήσεις, που σημαίνει ότι έχουν ένα ε, πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους προμηθευτές. Έχουν εξαιρετικές δηλαδή συνθήκες χρηματοδότησης που δεν μπορούν να προσφέρουν οι Ευρωπαίοι που πειθαρχούν στους κανόνες του ΟΣΑ. Ε, συγγνώμη, του ΟΕ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά αποτελούν ένα μεγάλο μειονέκτημα για την ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα, το πιο σημαντικό. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει η βιομηχανία μας αυτή να παραμείνει σε ηγετικό ρόλο. Η UNIFE εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ετοιμάσει ε, μια επίσημη έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μετά από την ε, έκθεση πρωτοβουλίας της ε, κυρίας Μαρτίνα Βέρνερ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό, τους κανόνες που ισχύουν και να εντοπίσουμε τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα συντονιστεί η ευρωπαϊκή αγορά για να είναι πιο ανταγωνιστική. Πρώτον, η προσφορά. Πρέπει να παράγουμε τα καλύτερα δυνατόν προϊόντα της αγοράς για να μπορούμε να τα εξάγουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ενισχύοντας την έρευνα και την ανάπτυξη και τον ορίζοντα 2020 και το shift to rail, πράγματα που το 2014 έγιναν πραγματικότητα χάρη στη στήριξη της Επιτροπής σας. Έρευνα και ανάπτυξη επίσης ε, για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συστάδες επιχειρήσεων, τα κλάστες. και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιοτεχνίες και τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, θα έπρεπε να βελτιώσουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε δύο σημαντικά πράγματα μπροστά μας. Την αναθεώρηση των κανόνων που χρειάζονται από τους προμηθευτές και από τους πελάτες και Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να ενισχύσει την ικανότητά μας στην εξαγωγική και να βελτιωθεί η πρόσβασή μας στις αγορές. Είτε πρόκειται για την Κίνα, είτε πρόκειται για την Ιαπωνία. Ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη δικιά σας στήριξη στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα και την, Ιαπωνία που είναι πολύ ευαίσθητες. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα μας και θέλουμε να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά έργα, όργανα και να υποφεληθούμε και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τις προτάσεις μας θα τις βρείτε και μέσα στο έγγραφο αυτό το οποίο σας έχουμε μοιράσει και είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και όλη την Επιτροπή σας που με προσκαλέσατε. Και ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα την Ευρωβουλευτή την κυρία Βέρνερ και τη δουλειά που έχει κάνει πάνω σε αυτό τον ε, τομέα, τον τόσο σημαντικό για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. κύριε Φίλιπ Σιτροέν για την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σας εισήγηση στην αρχή της συνεδρίας της Επιτροπής και τώρα να περάσουμε στην δεύτερη ομιλία. Ο ομιλητής μας είναι ο κύριος Ζαν Βεργιέρ. Εάν θέλατε κι εσείς, χωρίς να σας χρονομετρήσουμε και γι' αυτό, να πείτε λίγα λόγια για να συστηθείτε. Παρακαλώ συστηθείτε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βέρνερ, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Καταρχά σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή σα να σα μιλήσω. Είναι και τιμή μου και μεγάλη μου χαρά. Είμαι και Γάλλος πολίτης. Πριν από πάρα πολλά χρόνια γεννήθηκα στον παρά τη Γαλλία. Η πρώτη μου επαγγελματική σταδιοδρομία ήταν στον χώρο της Βιομηχανία στη Siemens. Κάποια χρόνια στη Γερμανία και μετά κατά κύριο λόγο στη Γαλλία σε τρεις ε, τομείς, στους αυτοματισμούς της βιομηχανίας, ε, την βιομηχανία μετά τις, και μετά στις μεταφορές, όπου ήμουν αναπληρωτής διευθυντής της κινητικότητας της Siemens για τη Γαλλία. Το 2008 ξεκίνησα μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία και έγινα σύμβουλος του πόλου καινοτομία, ε, ανταγωνιστικότητας iTrans, που ουσιαστικά δραστηριοποιείται στην Πικαρδία και στο Νορπάντε Καλέ, με ιδιαίτερη έμφαση στις υδροδρομικές μεταφορές. Με προσκαλέσατε εδώ ως πρόσωπο του δικτύου ΕΡΣΥ, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για, τις, ε, για τους κεντρωτικούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκε από την ε, iTrans. Και από ό,τι βλέπω ξεκίνησε και το χρονόμετρο. Το δίκτυο αυτό, το βλέπετε και στο χάρτη, δημιουργήθηκε βήμα το βήμα και χρονιά τα χρονιά. Είμαστε τώρα 10 συγκεντρωτικοί μηχανισμοί, σχηματισμοί από 10 διαφορετικέ χώρε με 7 διαφορετικέ γλώσσε, κάτι που δεν είναι καθόλου απλό. Και προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε φορεί από διαφορετικέ χώρε που έχουν ομοιότητε μεταξύ του ομοιότητε. βέβαια τίποτα δεν είναι παρομοιότυπο μεταξύ των διαφορών κρατών μελών, αλλά υπάρχουν ομοιότητε και στους στόχου και στο τι παθιάζει τον καθένα και τι όχι. Πριν προχωρήσω, να σταθώ στον όρο κλάστερ, συγκεντρωτικό σχηματισμό, ένα όρο που χρησιμοποιείται ευρέω στι Βρυξέλλε κυρίω. Αλλά θα ήθελα με τη συμφωνία σα να σταθώ στον ορισμό κλάστερ αρχικά από τον Μάικλ ε, Πόρτερ το 1980 ε, στο Harvard Business School δημιουργήθηκε ο όρος αυτός και είπε ότι Cluster είναι μια ομάδα επιχειρήσεων εταιριών, ε, θεσμικών φορέων που βρίσκονται στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές και διασυνδέονται με σχέσεις αλληλεξάρτησης για, ένα παρόμοιο, για μια παρόμοια ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών. Βεβαίω είναι πολύ γενικόλογοι και αυτοί, πολύ γενικόλογος αυτός ο ορισμός, αλλά υπάρχουν τρεις λέξεις κλειδιά. Πρώτα απ' όλα γεωγραφική περιοχή, ε, επικράτεια. Ε, ήδη αυτό είναι μια πολύ σημαντική έννοια, διότι υπονοεί την, ε, τον πολιτισμό, την ιστορία, έναν ιστό κοινωνικό και ανθρώπων, σχέσει αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων. Και βεβαίω εδώ παίζει ένα ρόλο και το διαδικτύο. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι η αλληλεξάρτηση. Υπάρχουν διαφορετικέ μορφέ αλληλεπίδραση ε, στα πλαίσια ενό ε, κλάστερ, ενό κεντρωτικού σχηματισμού. Μπορεί να είναι μια σχέση μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Μπορεί να είναι κάτι που σχετίζεται με την ε, εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων, ειδικών γνώσεων. Ή μια εταιρική σχέση των τομέα των επιχειρήσεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες εθνικές, περιφερειακές, πολιτικές αλλά και προσωπικές πρωτοβουλίες. Ε, μερικά παραδείγματα στην Ιταλία. Ε, υπάρχει μια τάση διοργάνωσης των μικρομεσαίων εταιριών σε κλάστερ και δύο σε εθνικό, σε επίπεδο για τις μεταφορές πάνω απ' όλα. Και στη Γερμανία δύο ειδών πρωτοβουλίες, το Go Cluster με με τα and Cluster επίσης μια δεύτερη πρωτοβουλία με τις 15 κορυφαίες ε, συγκεντρώσεις επιχειρήσεων και στην Γαλλία για την ανταγωνιστικότητα εδώ και 10 χρόνια υπάρχει μια δραστηριότητα από τον πόλο ανταγωνιστικότητας που με διαφορετικές εκλογικές ευκαιρίες έχει οικοδομήσει τους συγκεντρωτικούς σχηματισμούς στην Ισπανία από το 2007 υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται ARIES με σημαντικά κλάστερ ε, στην Καταλωνία κυρίως και θυμάμαι να έχω πάει στη Βαρσοβία, στο Υπουργείο Οικονομικών το 2013 να εξηγώ τι είναι η πολιτική των κλάστερ και η Πολωνία έχει πλέον και, και αυτή η πολιτική κλάστερ, οπότε είναι και αυτή μία ε, από τους εταιρείε μας. Στην Σουηδία ε, ένας από τους μαθητές του κυρίου Πόρτερ στο, του, καθηγητά, του καθηγητή Πόρτερ στο Χάρβαρντ ε, εισήγαγε και εκεί την πολιτική των κλάστερ. Τώρα, για τους στόχους του πόλου ανταγωνιστικότητας προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε ανθρώπους που έχουν ομοιότητες μεταξύ τους. Τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε προγράμματα συνεργασία για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Για να το εξηγήσω αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλέ φορέ το συγκρίνω με του καταλήτε τη χημικές αντιδράση. Στι χημικέ αντιδράσει, ένα καταλήτη δεν συμμετέχει ακριβώ στην ίδια την αντίδραση, αλλά χωρί τη δική του ε, δεν ξεκινάει η χημική αντίδραση. Αυτό θέλαμε κι εμεί να έχουμε ανθρώπου από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα για να συγκεντρωθούμε και να συνεργαστούμε για κοινά προγράμματα. Επιθυμούμε, και αυτή είναι η καθημερινή μα εργασία, μαζί με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει συνοδεύουμε στην οριμότητα, να ασχοληθούμε από το στάδιο των προμηθευτών σε επίπεδο συνεργασία και να συνοδεύσουμε τι εταιρείε στην στρατηγική ε, του ορίμανση, δηλαδή την ανάπτυξη μια στρατηγική ε, τη ίδια του τη ανάπτυξη και με δικό του χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων. Επίση, θέλουμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κοινοτομία και ανάπτυξη να εκφραστούν σε νέε υπηρεσίε στην ε, αγορά, βελτιωμένε και στόχο μα δεν είναι να είμαστε απλώ ένα κλαμπ ε, τη ελίτ των εταίρων, αλλά να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Εάν δούμε τι μορφή έχουν χαρακτηριστικά τα μέλη μας από κλάστερ, θα, θα δούμε ότι 42% μέσος όρος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί γιατί η προτεραιότητά μα ε, είναι όχι απλώ ο αριθμό των επιχειρήσεων που θέλουμε να συγκεντρώσουμε, αλλά και τι ανάγκη έχουν αυτέ οι επιχειρήσει να βοηθηθούν. Επίση είναι το πόσο ευάλωτε είναι και το πόσο κινητικέ. Είναι εταιρείε ε, εξαιρετικά καινοτόμε, ευέλικτε και σε θέση ε, να υποφεληθούν από τη δική μα στήριξη. Γρήγορα είδαμε ότι η δουλειά μα μπορεί να είναι χρήσιμη για την Ευρώπη εφόσον μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Η πεποίθηση αυτή και για μας και για τα μέλη μας είχε πραγματικά προστιθέμενη αξία ώστε να δημιουργήσουμε και αυτή την ε, πολιτική διασυγκεντρωτικών σχηματισμών για να έχουμε πρόσβαση σε νέες ειδικές γνώσεις, σε νέα εμπειρογνωμοσύνη. Ε, μπορέσαμε έτσι να υποφεληθούμε από το βλέμμα άλλων ε, πολιτισμών στο ίδιο θέμα Έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ιδίω για τι τεχνολογίε των σιδηροδρόμων, όπου τα ίδια πράγματα, εφόσον τα δούμε από μια διαφορετική σκοπιά από τη μια χώρα στην άλλη, καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα, πλουσιότερα. Ε, θέλουμε επίση να έχουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, ω προ τη διαχείριση, του ανθρώπινου πόρου, τι διαδικασίε που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίση, μαζί θέλουμε να αναπτύσσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, γνωρίζοντας ότι έχουμε μία βάση μελών και εταίρων που εμπιστεύονται οι μεν δε και γνωρίζονται καλά και από να αναπτύσσουμε δραστηριότητε στι αγορέ στόχου. Έτσι μπορούμε να διευρύνουμε την αγορά για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη, κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρω και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, για την ε, Ευρώπη των σιδηροδρόμων ε, υπάρχει μια μεγάλη προστιθέμενη αξία από πλευρά μα και εδώ θα, προσ... θα σταθώ σε ένα στοιχείο ιστορία. Ξέρετε ότι η βιομηχανία των σιδηροδρόμων πάντοτε είχε στρατηγική σημασία. Αυτό φάνηκε και στην ηθική επικράτεια του κάθε κράτου, αφού το σύνολο της προστιθέμενης αξίας αφορά τις πρωτεσίλες, τις ράγες, ε, τα υλικά, από όλα τα στάδια της εθνικής παραγωγής. Έπειτα ήρθε και η Ευρώπη να προσθεθεί σε αυτό και η αγορά άνοιξε σταδιακά. Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει ανοίξει ολοκληρωτικά, υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά άνοιξε και στην βιομηχανία των σιδηροδρόμων, το ξέρω Φιλίπ καλύτερα και από μένα, ε, υπήρξαν πολλές συγκεντρώσεις, συγχωνεύσεις, ε, εξαγορές και μεγάλες ευκαιρίες για τους μεγάλους πρωταθλητές της ε, βιομηχανίας των σιδηροδρόμων. Για αυτούς που παράγουν εξοπλισμούς, αυτούς που παράγουν υλικά και κάποιες, μικρές, και κάποιες λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι προέκυψε μια νέα πρόκληση. Οι μεγάλες εταιρείες προφανώς πήγαν και επένδυσαν στις χώρες που είχαν υψηλή ανάπτυξη και είχαν δίκιο να το κάνουν αυτό. Εκεί δημιούργησαν προστιθέμενη αξία, βρήκαν και άλλη προστιθέμενη αξία εκεί που πήγαν με τις ειδικέ γνώσει που του προσφέρθηκαν και ε, επίση, οι επενδυτέ, ιδίω τη Ασία, άρχισαν να έρχονται στην Ευρώπη για να επενδύσουν και να αναζητήσουν τεχνογνωσία. Η προστιθέμενη αξία των εθνικών κρατών κινδυνεύει να μετατοπιστεί για αυτό το λόγο. Ξέρουμε ότι δεν είναι ε, ε, δυνατόν να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην μηχανή των εξοπλισμών χωρίς να έχουμε μεγάλες εταιρείε και να έχουμε απλώς ένα ιστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που να είναι ισχυρές και καινοτόμε, αν δεν έχουν ε, τα ανάλογα εργαστήρια για τις μεγάλες μας έρευνες. Εδώ θα πρέπει η Ευρώπη να διατηρήσει την αξία της, κατά την απόψή μας. Υπάρχουν εδώ κάποιες μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι κάπως ευθύς η μεγάλη διαγωνισμοί με τα προγράμματα πλαίσιο και τον ορίζοντα 2020 λόγου χάρη είναι περίπου μη προσβάσιμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε κάτω μέλος, κάθε χρόνο καταρτίζει ένα κατάλογο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συμμετάσχει. Εάν δούμε κατά τι έχει συμβεί θα δούμε ότι κυρίως υπάρχουν ε, σύμβουλοι, consultants και πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πετυχαίνουν κάτι. Η διαδικασία είναι μακρά, ε, χρονοβόρα, ε, κοπιαστική και δαπανηρή. Αλλά υπάρχουν και καλά νέα. Ήδη με τη UNIFE έχουμε συνεργαστεί, καθώς και με τους ε, ε, μεγάλους πρωταγωνιστές της Shift Rail ε, για να έχουμε μια μεγάλη χαρτογράφηση των σπουδών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 100 από αυτές μπορούν σήμερα και είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι και να συμμετέχουν σε όλα αυτά. Αλλά ήδη από το 2013 έχουμε ξεκινήσει την ε, έρευνα για να δούμε τι θα γίνει με τις πρώτες προκηρύξεις της Shift Rail τις ερχόμενες εβδομάδες. Έχουμε αισιόδοξη προοπτική για όλα αυτά. Επίση, για το μέλλον των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, ε, μια άλλη καλή είδηση είναι αυτό που γίνεται. Και αν δούμε και τι δραστηριότητε ω προ την πολιτική των κλάστερ στην Ευρώπη, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πολλέ συγκριτικέ αξιολογήσει, ε, πολλά παράσημα αριστεία και αντιμετώπιση προκλήσεων, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί διαγωνισμοί για προγράμματα που σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν τα κλάστερ ω. έχουν. Μερικά παραδείγματα. Υπήρξε διαγωνισμός κόσμε και τώρα θα επιταχύνω που σκοπό είχε να διαλέξει 8 προγράμματα από 60 προτάσεις 80.000 ευρώ μεταξύ 5 εταίρων για 5 χρόνια δεν ήταν στο ύψος των αναγκών αλλά θα πρέπει τα πράγματα να βελτιωθούν. Το ίδιο και για το εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εδώ υπάρχουν καλέ ειδήσει, αλλά ένα ποσοστό επιτυχίας αρκετά χαμηλό, που δεν, περίπου 20%, που δεν είναι πολύ ε, δεν είναι κάτι που δίνει κινήτα. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς στο, ως Ευρωκοινοβούλιο, ιδίω η Επιτροπή σας. Να βεβαιωθείτε για την ευστοχία και την ε, καλή ε, επίδοση των κλάστερ, να δώσετε κίνητα στα κατημέλη για να προβλέψουν μια διαρκή βιώσιμη πολιτική για τα κλάστερ, κάτι που δεν ισχύει ακόμη. Να υπάρχει ένα σύστημα κρατικών χρηματοδοτήσεων δημόσιων γιατί μιλάμε για υπηρεσίε κοινή ωφελία κάποιε φορέ και να βεβαιωνόμαστε ότι ο κανόνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 20% κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει πραγματικά να γίνεται σεβαστό. Εδώ πρέπει να γίνεται ένα έλεγχο πολύ σοβαρό. Και τέλο, πάνω απ' όλα, να υπάρξει λιγότερη περιπλοκότητα. Αυτό το χρειαζόμαστε όλοι. Και επιτρέψτε μου να κλείσω στα γερμανικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Προσπάθησα να συνοψίσω σε λίγα λόγια κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, κάποια μηνύματα. Είμαστε στη διάθεσή σας στη συνέχεια. Και προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βεριέ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Το ότι αλλάξατε γλώσσα δεν σημαίνει ότι έχετε άλλα 10 λεπτά χρόνο ομιλίας. Ωστόσο ήταν ωραίο που είπατε λίγα λόγια στα γερμανικά στο τέλος της παρέμβασής σας. Η συγκήτριά μας, η κυρία Βέρνερ, ε, θα ήθελα να πάρει το λόγο. Τρία λεπτά αρκούν. Τρισήμιση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιτροέν, κύριε Βεριέ, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τον σιδηροδρομικό τομέα και που έχουμε εδώ τους δύο εμπειρογνώμονες για να σχηματίσουμε μια εικόνα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σιδηροδρομικός τομέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορέσατε να παρευρεθείτε. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε ένα παρόμοιο θέμα στην Ολομέλεια, την κρίση στην βιομηχανία Χάλιβα και νομίζω ότι τα δύο αυτά θέματα συνδέονται μεταξύ τους και στον τομέα του Χάλιβα και στον σιδηροδρομικό τομέα ε, μας ανησυχεί η στάση της Κίνας. Το 2002 είχαμε το πρώτο μετρό από την Κίνα. Σήμερα κάθε δεύτερο τρένο μετρό προέρχεται από την Κίνα. Και κύριε ε, είπατε ότι ε, η μεγαλύτερη βιομηχανία συνδρομικού υλικού ε, είναι κινέζικη και επιδοτείται αδρά από το κράτος. Εδώ και αρκετό χρόνο. Ε, αυτός ο ε, κινέζικος κατασκευαστής ε, προσπαθεί να επικρατήσει και στην διεθνή αγορά. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνδέονται όμως με το σιδηροδρομικό τομέα και γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα το ψήφισμα, διότι το ψήφισμα αναφέρεται σε θέματα που συχνά παραβλέπονται διότι θεωρούμε ότι είναι θέμα μεταφορών αλλά είναι εξίσου θέμα βιομηχανίας. Ε, και μια καλή συνδρομική βιομηχανία αποτελεί την βάση για ανάπτυξη και για μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν υπάρχουν εδώ εύκολες λύσεις. Ε, χρειάζεται μια δέσμη μέτρων και στο ψήφισμα σχεδιάζω να θέσω όλες αυτές τις απόψεις, ε, κάποιες λέξεις κλειδιά, το shift to rail που αναφέρατε, ε, την πρόωθηση της καινοτομίας με έμφαση στην ψηφιοποίηση, προώθηση της καλύτερης πρόσβασης στην αγορά, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, καλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση ε, θέμα είναι και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τέλος εξίσου σημαντικό τα κοινά πρότυπα στην ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια εικόνα σχετικά με την κατάσταση στον τομέα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε έναν πιο καινοτόμο σιδηροδρομικό τομέα. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνεργατικοί σχηματισμοί ε, είναι καλά παραδείγματα του πώς ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα το σχέδιο ψηφίσματος. Σκοπεύω να το ολοκληρώσω μέχρι τις 27 Ιανουαρίου για να μεταφραστεί. Στις 22 Ιανουαρίου θα συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή. Η 25 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και 7 Απριλίου έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Εάν έχετε προτάσεις, ε, επιθυμίες για τροποποίηση του κειμένου κλπ. Παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Ε, καταρχάς όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε και άλλες ερωτήσεις ε, στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, πρόκειται για προφορική ερώτηση που ε, θα ακολουθηθεί από ένα ψήφισμα πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία η συζήτηση. Η κυρία Φρανσουάς Κροστέτ αντικαθιστά την κυρία Μοράνο από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η κυρία Μοράνο που είναι σκέδωση συζητήτρια για το ΕΛΚ λείπει και επειδή και ο κύριος Καρίνς είναι ο συντονιστής μας και εκείνος λείπει, θα πάρω εγώ το λόγο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους δύο εμπρογνώμονες με τις ε, πραγματικά ε, συναρπαστικές ομιλίες τους. Μας είπαν πόσο επίγει να κάνουμε κάτι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουμε την βιομηχανία εξοπλισμού των σιδηροδρόμων. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τη δουλειά της και θα είμαστε στο πλευρό της Γιατί αυτό που προέχει είναι να στηρίξουμε αυτή τη βιομηχανία μα που περνάει δύσκολε στιγμέ. Η ανταγωνιστικότητα τη πλήτεται από τον έντονο ανταγωνισμό από τρίτε χώρε. Κυρίω, μα το είπε ο κύριο Σιτροέν, καταλάβαμε ότι η Ασία διαρκώ φτάνει πιο κοντά στην Ευρώπη, κυρίω ό,τι αφορά του εξοπλισμού των σιδηροδρόμων, και αυτό μα ανησυχεί. Ωστόσο, αυτό το εξήγησαν οι δύο ομιλητέ μα, αλλά και η συγγετριά μας, η βιομηχανία των σιδηροδρόμων είναι στατηγική σημασίας. Είπαμε ότι 400.000 άτομα στην Ευρώπη απασχολούνται σε αυτή τη βιομηχανία. Πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη. Ε, και ιδιαίτερα ποικιλόμορφη. Είναι ενό είδου ε, αλυσίδα υπεργολαβία. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο μεγάλε εταιρείε, αλλά πάρα πολλέ μικρομεσαίε που συνεργάζονται με πάρα πολλούς ε, παραγωγούς εξοπλισμών και παρόχους υπηρεσιών. Και επίσης, μας εξηγήθηκε και αυτό, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στον τομέα αυτό. Στο επίπεδο όχι απλώς της Ευρώπης, αλλά διεθνώς. Η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Για να μην μπορεί να κατακτήσει μια σημαντικότερη θέση πρωτιάς της ε, στα μερίδια της νέας αγοράς, είτε στην Ασία, τη Μέση Ανατολή ή στην Αφρική. Βλέπουμε πόσο αυτές οι προκλήσεις είναι καθοριστικές. Μας είπε και η κυρία Βέρνερ και το συζητήσαμε με αφορμή την κρίση στη Χαλιβουργία. Είναι ένα μέσο για να ανταποκριθούμε στι ανάγκε αυτή τη κρίση, στηρίζοντα με κάθε τίμημα την ε, βιομηχανία των συντηροδρόμων. Είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε τι προσπαθίε μα σε αυτό το στόχο και γι' αυτό στρέφουμε και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απολύτω αναγκαίο να αναλάβετε σοβαρή δράση για να επιτρέψετε σε αυτή τη βιομηχανία να ανταγωνίζεται ισότιμα ε, τι τρίτε χώρε, Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν αρκεί να τα λέμε μόνο, πρέπει και να δράσουμε. Εάν λοιπόν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχει ένα βιώσιμο μέλλον αυτή η βιομηχανία μα ή η βιομηχανία των συνδροδρόμων στην Ευρώπη, για να κατακτήσει νέα μερίδια αγορά στην Ευρώπη, τώρα πρέπει να δράσουμε. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ε, στηρίξουμε, να ενισχύσουμε του πρωταθλητέ μα αυτέ τι πρωτιέ του συντροδρόμου θέλουμε να τι διατηρήσουμε. Αλλά όπω είπε και ο κύριο Βεργέ, ε, πρέπει να δώσουμε πρόσβαση ε, πιο εύκολη πρόσβαση, άνετη πρόσβαση στις μικρομεσαίε μα. Η ευρωπαϊκή λοιπόν απόκριση πρέπει να είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση των επενδύσεων υπέρ τη κοινοτομίας και της έρευνας μέσω των clusters. Πολύ σωστά μας εξηγήθηκε αυτό. Αυτό θα είναι η προσταθέμενη αξία τη δική μα βιομηχανία και σύντομα ολοκληρώνω. Ε, από την άλλη, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία εμπορική μας άμυνας και τους κανόνες, τους κανόνες που δεν θα πρέπει να είναι αφελείς, αφελείς ως προς την ε, ε, απόδοση των ε, δημόσιων προμηθειών. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες, να διευκολύνουμε τους εργαζομένους αυτών των, αυτού του χώρου με ιδιαίτερα προσόντα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η Ευρώπη δεν θα καταλήψει αυτή τη βιομηχανία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία μου, για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Ρικέ. Shadow Rapporteur. Σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα τα πω σύντομα για να πω ποιες είναι οι απόψεις μας, ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιες είναι οι ελπίδες που έχουμε. Περιορισμούς έχει ο κλάδος εξαιτίας της ίδιας της δομής του. Αναφέρθηκε και ο κύριος Σιτρά την αναδιάρθρωση του τομέα που δεν φτάνει. Ο ανταγωνισμός είναι διεθνής, δεν υπάρχει συνεργασία μέσα στην Ευρώπη και ούτε αρκετή αναδιάρθρωση στις ε, μεγάλες επιχειρήσεις συναρμολόγησης. Οι επιχειρήσεις μας υποφέρουν, δεν είναι καλά οργανωμένες, πιέζονται, υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά τεχνολογίας και δεν έχουν πρόσβαση σε ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα για τα οποία ανησυχούμε. Τώρα στο ιστορικό υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα και διεθνώς υπάρχουν μεγάλοι γίγαντες, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δηλαδή αυξάνεται. Και υπάρχει και το θέμα της μετεγκατάστασης, όταν οι επιχειρήσεις μας ε, κερδίζουν ε, αγορές πρέπει να ε, μεταφέρονται εκεί και έχουμε τέτοια παραδείγματα πρόσφατα. Η μεταφορά τεχνολογίας επίσης όπως των βαβαρδιστικών που πήγε στην Κίνα. Στο εσωτερικό πάντως της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οικονομική κρίση και έλλειμμα ρευστότητα στις χώρες μας. Κατακαιρματισμός επίσης στην αγορά. Κατακαιρματισμός και στον χώρο μέσα στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη. Τέλος, προχωρούν και οι άλλοι τρόποι μεταφοράς. Οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές κερδίζουν έδαφος πω το υπενθυμίσατε κι εσείς, εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι στον κόσμο με 46% με πραγματικά προϊόντα εχμής και όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογία επίσης. Αλλά πρέπει και στην τυποποίηση να κάνουμε πρόοδους. Και η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να προχωρήσει στα πλαίσια του shift to rail. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πρόσβαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλα αυτά. Οι ισοδρομικές μεταφορές είναι αυτές που προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον και χρησιμοποιούν και λιγότερα ορυκτά για την, ε, ως ενέργεια. Πρέπει να μειωθεί και το κόστος και νομίζω το τέταρτο πακέτο σειροδρόμων μπορεί να βοηθήσει πρέπει να επωφεληθούμε και από την ψηφιοποίηση, να ανοίξουμε τις αγορές, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των συνοδρόμων ως τρόπος μεταφοράς, αλλά όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών είμαι μάλλον απεσιόδοξος, αλλά χρειάζεται αναδιάρθρωση για να φτάσουμε να έχουμε το Airbus στους σιδηροδρόμους. Επίσης, πρέπει να υπάρχει υπεργολαβία σταθερά και να βελτιώσουμε και τον ε, ανταγωνισμό τηρώντας την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Ώστε ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, ο αντίστοιχος κλάδος να πληρώνει. Επίσης, στην Ευρώπη να ενισχύσουμε και το τροχαίο υλικό στους σιδηροδρόμους. Είναι ένα θέμα που πρέπει να θέσουμε επιτάπητος. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τους Ιάπωνες και τους Κινέζους να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Η κυρία Κάπελ είναι η επόμενη ομιλήτρια με μέρου της ομάδας ENF. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιτρόεν, κύριε Βεριέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε για το σημαντικό αυτό θέμα των ε, κατασκευαστών ε, σιδηροδρομικού υλικού της Ευρώπης. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει της, ε, του ενδιαφέροντος που το αξίζει στο κοινό. Υπόθηκε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδηροδρομικού υλικού είναι πολύ σημαντική βιομηχανία ε, στην Ευρώπη ε, κατέχει το 46% του, της διεθνούς αγοράς και το πρόγραμμα Shift to Rail είναι πολύ σημαντικό. Χρηματοδοτείται με 920 εκατομμύρια ευρώ, το ίμιση των οποίων προέρχεται από το ορίζον. Και υπό το φως της παρούσας διάσκεψης COP21 ε, πρέπει να αναφέρουμε ότι η βιομηχανία σιδηροδρομικού υλικού έχει τις ε, χαμηλότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από τις βιομηχανίες μεταφορών της Ευρώπης. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό να βρίσκεται στο θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέδια στο Στρασβούργο συζητήσαμε την κρίση στον τομέα του Χάλιβα. Είναι υψηλές οι τιμές, βρισκόμαστε σε κακή οικονομική συγκύρια και ε, έχουμε πλημμυρίσει από προϊόντα από τρίτες χώρες. Επίσης, προβληματική είναι η περιορισμένη πρόσβαση της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας συνδρομικού υλικού ε, στην Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε καλές διαπραγματεύσεις. ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά. Και άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ε, Κίνας. Η κινέζικη εταιρεία CCRS ε, με 31 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση έχει το μέγεθος των δύο τρίτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να έχει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε αυτό απέναντι στην Κομισιόν, το θέμα δηλαδή του δικαίου ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ε, thank you, ε, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαν. Θα ήθελα να επικροτήσω αυτά που είπε η συγγήτριά μας ε, η Μαρτίνα Βέρνερ είναι σημαντικό το θέμα της ψηφιοποίησης. Ε, στην, στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε με την αποστολή για την Κίνα το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και του ντάμπινγκ στον τομέα του χάλιβα. Το βλέπουμε αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ακριβώς ε, δείχνει την ανάγκη να έχουμε ενιαία βιομηχανική πολιτική, να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές του θέματος. Όσον αφορά τα, τους συνεργατικούς ε, σχηματισμούς, ε, τα κλάστερ, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Έγινε πολλή δουλειά με τα διαστρωτικά ταμεία ώστε ε, στα συνεργατικά δίκτυα να έχουμε άμεσα αποτελέσματα ώστε τα αποτελέσματα που επιτυχάνονται σε έναν βιομηχανικό τομέα να μεταφέρονται σε άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω και στους δυο σας. Κυρίως για τον κύριο Σιτρόεν στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε στους μηχανισμούς, τους διαθέσιμους χρηματοδότησης και ολόκληρο τον κλάδο και για τους τέσσερις τομείς που μας αναφέρατε. Είμαι περίεργος, λοιπόν. Θέλω να ξέρω πώς ο σιδηροδρομικός κλάδος δέχεται και χρησιμοποιεί το σχέδιο Juncker. Έχετε ήδη κάποια προγράμματα που να έχετε υποβάλει και σε τι βαθμό αφορούν τον καθένα από τους τέσσερις τομείς τους οποίους αναφερθήκατε. Και για τον άλλο μας συζητητή, στον τομέα της καινοτομίας και της ανάπτυξης και της έρευνας, οι πολιτικές των κλάστερς συμπεριλαμβάνουν και την δυνατότητα να συμπληρωθούν από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το σχέδιο Juncker. Υπάρχει συνδυασμός χρηματοδότησης. Το σχέδιο Juncker έχει αξιοπιστία και γίνεται αποδεκτό από τον κλάδο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, Θέλω να απευθυνθώ στην Επιτροπή, την Γενική Διεύθυνση Growth, η κυρία Ιωάννα Κρυπόφσκα. Σωστά. Αν έχετε κι εσείς απαντήσεις ή αν έχετε κάτι να προσθέσετε στη συζήτησή μας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσω πολλά στη συζήτησή σας και να την κάνω πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι ήδη είναι. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να συμμετάσχει στην τόσο σημαντική αυτή συζήτηση. Χαίρομαστε πολύ για την πρωτοβουλία της κυρίας Βέρνερ για έκθεση όσον αφορά τον, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας του δρομικού υλικού και σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια. Πολλοί ομιλητές ήδη αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει ο κλάδος αυτός για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος Προμήθειας για μας είναι ζωτικής σημασίας και ανάπτυξή του είναι κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως υπάρχουν όλες οι προκλήσεις τις οποίες αναφερθήκατε Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να αναπτυχθεί παρετέρω, ότι πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση ισότιμη στη χρηματοδότηση, δίκαιος ανταγωνισμός και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις και τα προβλήματα. Αναφερθήκατε και στην συνεργασία και υπάρχουν πολλές καλές λύσεις και εσείς αναφέρατε δύο. Το τέταρτο σερνομικό πακέτο για παράδειγμα, το οποίο θα έπρεπε να οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Ελπίζουμε να εγκριθεί σύντομα, να μην υπάρχουν ούτε τεχνικές ούτε νομικές ε, δυσκολίες και κολλήματα. Αναφερθήκατε και στην πρωτοβουλία Shift to Rail. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μας βοηθήσει να έχουμε πανευρωπαϊκές λύσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος του κλάδου προμήθειας δρομικού υλικού παγκοσμίω. Υπάρχουν ήδη εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή που αναπτύσσονται αυτή την εποχή και σε συνεργασία μαζί σας και με τον κλάδο θα προσφέρουμε τη στήριξή μας. Θα προσφέρουμε τη στήριξή μας και στην κυρία Βέρνερ για την έκθεση την οποία ετοιμάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα, στρέφομαι στους ομιλητές μας ο κύριος Σιτροέν και ο κύριος Βεριέ. Παρακαλώ να απαντήσουν και να λύσουν διάφορες απορίες που εκφράστηκαν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τους ευρωβουλευτές. Έχω την εντύπωση ότι κατάλαβαν πολύ καλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας κίνδυνοι που προέρχονται από την Ασία παρόλο που ο κλάδος μας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές όσο καλύτερα μπορεί. Σημείωσα διάφορα σημεία εδώ για την έρευνα και την καινοτομία συνεχίζουμε με δυναμισμό για το shift to rail ξέρουμε ότι είναι μια εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα και Θέλουμε όλα αυτά να αρχίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς που προβλέπονται. Το όλο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η εσωτερική αγορά να προχωρήσει. Αναφερθήκαμε στο τέταρτο πακέτο, αλλά υπάρχει και το θέμα των ε, δημοσίων ε, των διαγωνισμών για δημόσιες προμήθειες. Και πολύ συχνά ακούμε για ισότιμες συνθήκες εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά όταν υπάρχει η Απωνία, η Κίνα και οι συμφωνίες όπως αυτές προβλέπονται στο TTIP έχουν σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε από τον ανταγωνισμό. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ορθάνυχτη την πόρτα μας ε, στις, ε, στους ξένους, αν και αυτοί δεν κάνουν το αντίστοιχο για τις δικές μας ε, επιχειρήσεις. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι χαίρομαι πολύ αν μπορώ να συνεργαστώ με την κυρία Βέρνερ για την έκθεσή της που είναι ζωτική σημασία για τον κλάδο μας. Κάτι τελευταίο θέλω να προσθέσω. Στον Ισπανό Ευρωβουλευτή που ρώτησε για το σχέδιο Juncker. Δεν σας κρύβω ότι προχωράμε σιγά σιγά στο συνδρομικό τομέα. Είτε πρόκειται για το τρένο υψηλή ταχύτητα, είτε για άλλα. Δύσκολα βρίσκουμε ιδιωτικέ επενδύσεις για τέτοιου είδου προγράμματα. Πολλές ελπίδες έχουμε για ένα πρόγραμμα που θα έχει να κάνει με το RTMS. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει λευκό καπνό. Τέλος πάντων δεν ε, έχουμε υπόψη μας να προχωρήσει πολύ η ιστορία των κλάστερς μέσω αυτού του ταμείου. Ευχαριστώ. Και τώρα να ζητήσω από τον κύριο Βεργέ να σχολιάσει και να απαντήσει. Και εγώ ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Οφείλω και εγώ μια απάντηση στον Ισπανό Ευρωβουλευτή. Σίγουρα υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις, όπως με την ενέργεια, αλλά δεν θα κάνω εδώ ανάπτυξη όλων των μεγάλων θεμάτων που αφορούν ε, τους υδροδρόμους. Υπάρχουν όμως τρεις. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και προστασία του περιβάλλοντος, Άρα σίγουρα υπάρχει ένα σκέλο που συνδέεται με την ενέργεια. Ένα άλλο τομέα είναι η καλύτερη χρήση των υποδομών και των εγκαταστάσεων. Και ο τρίτο τομέα είναι η ψηφιακή εξέλιξη και το πώ επηρεάζει του σιδηροδρόμου. Όλε μα οι εργασίε και στον επίπεδο των κλάστερ και στη συνεργασία μεταξύ μα είναι κάτι, το είπα και νωρίτερα, στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την DG και με τις εθνικές, με τις συνεργασία με εθνικούς φορείς και τις μεγάλες εταιρείες. Να προσθέσω επίσης, δεν το είπα προηγουμένως, καθένας από εμά στην δική του την ε, περιοχή συνεργάζεται με τις περιφερειακές αρχές για την υλοποίηση της Smart Specialization Strategy, ιδίως για την επιλογή των προτεραιοτήτων. Η δική μας πείρα ήταν ε, η πραγματική συμβολή στην περιφερειακή υλοποίηση αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τι παρατηρήσει και τι απαντήσει σα. Κυρία Μαρτίνα Βέρνερ, η συγκεκριά μα. μπορείτε να ανακεφαλαίωσετε τη συζήτηση, να συνοψίσετε ότι υπόθηκε και να μα πείτε τι θα γίνει στο μέλλον για την έκθεση αυτή κυρίω. Ναι κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιτροέν και κύριε Βεργέ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές και όσους συμμετείχαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο που ασχοληθήκαμε σήμερα αναλυτικά με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έτσι έχουμε καταλήξει στα βασικά θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ψήφισμα. Τη σημασία του συνδρομικού τομέα για την Ευρώπη, ε, καινοτομία, shift to rail, ε, πολιτικό ανταγωνισμού, συνθήκες ισονταγωνισμού, COP21 ε, πιθανότατα τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτά λοιπόν είναι θέματα στα οποία θα επικεντρωθούμε. Σίγουρα ε, θα μπορούσε να πει κανείς ε, πολύ περισσότερα. Το πρόβλημα είναι πώ θα τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά σε δύο σελίδες. Πάντως ε, με τα όσα ακούσαμε διαπιστώνω ότι όλοι σκεφτόμαστε περίπου με τον ίδιο τρόπο. Προσβλέπω λοιπόν στη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό το ψήφισμα αυτό, διότι όλοι πηγαίνουμε προ την ίδια κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι πολύ καλή και η συνεργασία μαζί σα Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εξέταση ε, του σχεδίου ψηφίσματος θα γίνει 22-23 Φεβρουαρίου. 25 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, δύο μέρες αργότερα δηλαδή. Ψηφοφορία στην Ήτρα, όπως είπατε και εσείς, στις 7 Απριλίου. Αυτό λοιπόν ήταν το χρονοδιάγραμμά μας. Ε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστήσω θερμά τους προσκεκλημένους μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορέσατε να παρευρεθείτε και οι δύο στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. We continue our meeting in... Συνεχίζουμε αμέσως τη συνεδρίασή μας γιατί έχουμε καθυστερήσει, στη μελέτη για την αποθήκευση ενέργειας. Τι σχεδιασμό στην αγορά χρειάζεται και τι κίνητρα νομοθεσίας από τον δόκτωρα Σέρχιο Γκάρτε για την βιώσιμη ποιότητα. Αυτό θα πει SQ. SQ Consult BV. Η μελέτη διεξήχθη από την Υπηρεσία Πολιτικής ε, κατά Αιτήματος της Επιτροπής Ήτρε με τίτλο, όπως είπα, αυτό που ανέφερα, η μελέτη θέλει να περιγράψει τι σχεδιασμό στην αγορά και τι νομοθετικέ ε, αλλαγέ χρειάζονται για να ε, υποθάλψουν αυτή την πολιτική και να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών αποθηκεύσης ενέργειας. Μόνο με τέτοιε τεχνολογίες θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να συμβάλλουμε του στόχους τη Ενεργειακή Ένωσης, δηλαδή την ασφάλεια της ε, προμήθειας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ε, καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην έρευνα και την απαλλαγή της οικονομίας από το χάλιβα, από τον Άντσακα, συγγνώμη. Ε, να ζητήσω από τον δόκτορα Ουγκάρτε να μας παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του και τη μελέτη για το θέμα αυτό. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Για δυστυχώς μόνον 10 λεπτά. Παρακαλώ, όχι παραπάνω. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα παραμείνω στα 10 λεπτά. Η μελέτη που θα σας παρουσιάσω μας ανατέθηκε από τον ε, τομέα πολιτικής Α. Τι σχεδιασμός αγοράς και τι κίνητρα χρειάζονται σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσουν να προωθήσουν την αποθήκευση της ενέργειας ε, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού ε, Συστήματος Ενέργειας. Θα διατρέξω πολύ σύντομα το πεδίο εφαρμογή ε, και τον στόχο. Ποια είναι η αξία της αποθήκευσης ενέργειας για το σύστημά μας, ε, ποια είναι η αξία της ε, αποθήκευσης ενέργειας, πώς συμβάλλει η αποθήκευση ενέργειας στην Ενεργειακή Ένωση. διότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ε, συζήτησης για την Ενεργειακή Ένωση. Κατόπιν ε, θα ασχοληθούμε με τις ε, μελλοντικές εξελίξεις, τα σημεία συμφόρησης και τις συστάσεις που συνδέονται με αυτές τις δυσκολίες, τα σημεία συμφόρησης. Ο στόχος, όπως ήδη υπόθηκε, είναι να σας βοηθήσουμε στην συζήτηση πώς μπορείτε να ταιριάξετε την αποθήκευση άνθακα μέσα στην όλη συζήτηση για την Ενεργειακή Ένωση. Στοχό είναι να προωθηθούν οι ενέργειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να ε, έχουμε μια οικονομία απειλαγμένη από τις ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και να έχουμε ασφάλεια τροφοδότηση. Έχουμε επικεντρωθεί σε 37 ερωτήσει. Ποια είναι η αξία τη αποθήκευση ενέργεια, ποιο είναι το κόστο των τεχνολογιών, πώ συμβάλλουν στην Ενεργειακή Ένωση και την απαλλαγή τη οικονομία από τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, έχουμε λοιπόν κατάλογο των ερωτήσεων. Ε, μπορείτε στο ευρετήριο της έκθεσής μας να βρείτε τις απαντήσεις. Ποια είναι λοιπόν η αξία της αποθήκευσης ενέργειας. Βλέπετε εδώ την αλυσίδα αξίας για την ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρώτα έχουμε τις πηγές ενέργειας, το, φυσικό αέριο, ε, ε, ε, κάψιμα κλπ. Κατόπιν έχουμε την παραγωγή ενέργεια, την μεταφορά μεταξύ διαφόρων περιφερειών, την διανομή και τέλος έχουμε τον τελικό καταναλωτή ο οποίος όπως γνωρίζουμε τώρα μπορεί να παράγει μόνο σε ηλεκτρική ενέργεια και έτσι να την αποθηκεύσει. Έχουμε δύο είδη αποθήκευσης ενέργειας. Ε, μεγάλης κλίμακας, ε, δηλαδή σκεφτείτε τεράστιες δεξαμενές ε, φυσικού αερίου, νερού, συμπιεσμένου, πεπιεσμένου αέρα στο υπέδαφος. Αυτό στην αλυσίδα αξίας ε, βοηθάει κυρίως τα πρώτα στάδια, την παραγωγή και την μεταφορά ενέργειας. Μετά ε, έχουμε ε, διάφορες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας σε μικρότερης κλίμακας. Κάτι που βοηθάει στην μεταφορά και την διανομή καθώς και τον τελικό καταναλωτή. Η αποθήκευση η ενέργειας μεγάλης κλίμακας ε, μπορεί να βοηθήσει την ε, ασφάλεια τροφοδοσίας, να διασφαλίσει την ασφάλεια ε, τροφοδοσίας σε περίπτωση για παράδειγμα που έχουμε λήψεις στην τροφοδοσία φυσικού αερίου κατόπιν κατά την παραγωγή είναι κάτι που βοηθάει στην απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές γιατί διότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγεται με αποβιώσιμες πηγές ενέργειας. εολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια κλπ. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια και να την διοθετεύσουμε ε, στο δίκτυο αργότερα, μπορούμε έτσι να αντικαταστήσουμε ε, άλλες πηγές ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια κλπ. Μπορεί κανείς να αποθηκεύει την ενέργεια όταν είναι ευθυνή και να την ε, καταναλώνει όταν είναι πιο ακριβή. Όσον αφορά την μεταφορά, η αποθήκευση ενέργειας ε, βοηθάει στη σταθεροποίηση του δικτύου. Έχουμε τώρα Περισσότερε βιώσιμε πηγέ ενέργεια, οι οποίε όμω εξαρτώνται από την ε, ηλιακή ακτινοβολία, από την ταχύτητα του ανέμου κλπ. Υπάρχουν ε, λοιπόν με τι βιώσιμε πηγέ ενέργεια ε, περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την σταθερότητα του δικτύου. Η αποθήκευση ενέργειας όμως βοηθάει να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι διακυμάνσει. και επίση, όσον αφορά την διανομή βλέπουμε ότι σε το, το χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα όταν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση για θέρμανση ή για κλιματισμό. Πάλι η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να μας ε, βοηθήσει και ε, επίσης τον τελικό καταναλωτή μπορεί να βοηθήσει διότι κάποιος που παράγει μόνο του την ενέργεια μπορεί να έχει και κάποια συσκευή αποθήκευσης της ενέργειας και να την καταναλώνει όποτε θέλει. Όσον αφορά την ε, οριμότητα των τεχνολογιών, ε, το πόσο έτοιμες είναι οι τεχνολογίες, ε, μου είπατε ότι έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου, ήδη, έχουν περάσει τα 5, οπότε σας αφήνω αυτή την διαφάνεια να τη μελετήσετε με την ησυχία σας αργότερα. Όσον αφορά τα θέματα πολιτικής, πράγματα που σας ενδιαφέρουν εσάς. Η αποθήκευση ενέργειας, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτήν, πώς, πώς μπορεί να συμβάλλει όμως στην Ενεργειακή Ένωση. Ε, ασφάλεια τροφοδοσίας. Ε, σκεφτείτε την αποθήκευση ε, φυσικού αερίου. Αυτό φυσικά ε, διασφαλίζει την τροφοδοσία σε περιοχές που εξαρτώνται από το φυσικό αέριο. Τι χώρες της Βαλτικής, η Βουλγαρία, η Φιλανδία εάν έχουν καλές εγκαταστάσεις αποθήκευσης ε, του φυσικού αερίου μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα που υπάρχουν και άλλα όσον αφορά την προμήθεια του φυσικού αερίου. Όσον αφορά την ολοκλήρωση, την ολοκλήρωση των αγορών ενεργείας. Η αποθήκευση ενέργειας είναι μία από τις λύσεις που είναι στη διάθεσή μας σήμερα ε, που παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία για να υπάρξει ολοκλήρωση της ε, αγοράς ενεργείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέθεσε μία έρευνα για την για το δυναμικό όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα χρηματοδοτούνται εργοστάσια παραγωγής ενέργειας για να υπάρχει σταθερότητα του δικτύου. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις. Ε, πρόκειται για αυτές τις λύσεις ευελιξίας ακριβώς και η αποθήκευση ενέργειας είναι μία από αυτές τις λύσεις. Είναι κάπως δαπανηρή, αλλά μακροπρόθεσμα ε, είναι μια ανταγωνιστική επιλογή. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, εδώ είναι αρκετά μικρός ο αντίκτυπος, διότι υπάρχουν απώλειες κατά την αποθήκευση. Ωστόσο, εάν αποθηκεύουμε την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό είναι καλό, διότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τον στόχο μας όσον αφορά την απαλλαγή της οικονομίας από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι δεν σπαταλάμε απλά την ενέργεια που παράγεται, μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε όταν την έχουμε ανάγκη. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ε, είναι επίσης η αποθήκευση της ενέργειας ένα παράγοντα που μπορεί να σταθεροποιήσει τις τιμές. Μπορούμε έτσι να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές ενέργειας. Το κόστος. γνωρίζετε ότι για τον ε, τελικό καταναλωτή υπάρχει ισοδυναμία δικτύου όσον αφορά τη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Η τιμή δηλαδή είναι ίση με το ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο του χρόνου. Θα επιτευχθεί ισοδυναμία δικτύου και για την αποθηκευμένη ενέργεια. Μαζί λοιπόν με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμα και αν είναι πιο ακριβές τεχνολογίες, θα έχουμε ισοδυναμία δικτύου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ε, η Γερμανία. Τα ευθύ e δίκτυα, τα έξυπνα δίκτυα, αν αυξάνεται ο αριθμός τους, όπως ε, και η ηλεκτροκινητικότητα. 40 δευτερόλεπτα μου απομένουν, έτσι. Ε, ας κοιτάξουμε λοιπόν ε, τα, τις ρυθμιστικές δυσκολίες. Βρίσκομαι στις δύο τελευταίες διαφάνειες. εάν ε, η Ευρώπη επιλέξει να χρησιμοποιήσει την αποθήκευση ενέργειας. Ε, τι θα γίνει. Η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κορέα και η Κίνα ηγούνται όσον αφορά τις έρευνες. Η Ευρώπη δυστυχώς ακολουθεί παρότι υπάρχουν ε, κάποια ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη, κάποιοι τομείς όπου βρισκόμαστε μπροστά από τους άλλους. Επίσης, όσον αφορά την αποθήκευση φυσικού αερίου, ε, έχουμε κάποιες μεγάλες δεξαμενές, αλλά οι χώρες της Βαλτικής, για παράδειγμα, η Βουλγαρία, εξαρτώνται από εξωτερική τροφοδοσία και υπάρχει εδώ έλλειψη διαφάνειας ε, στην αγορά και γι' αυτό δεν γίνεται επαρκής αποθήκευση φυσικού αερίου για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες ε, στην αγορά. Επίσης, η παραγωγή βιώσιμης ενέργειας αμείβονται επαρκώς στην Ευρώπη, δεν έχουν όμως καμία ευθύνη όσον αφορά την διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου. Τέταρτον, αναφέρθηκα και στην ευελιξία. Και τέλος, Υπάρχουν ε, προβλήματα όταν οι διαχειριστές των ε, δικτύων ε, δεν μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια διότι θα πρέπει αυτό να μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα του δικτύου. Και τέλος δεν έχουμε επίσης εγγύσεις για το τελικό καταναλωτή ακόμα. Και περνώ στην τελευταία διαφάνεια. Οι συστάσεις μας. Πάνω-πάνω βλέπετε την αλυσίδα τροφοδοσίας. Βλέπετε τα διάφορα στάδια. Βρήκαμε έξι δυσκολίες και έξι συστάσεις θέλουμε να υποβάλουμε στην Ευρώπη σε περίπτωση που θέλει να προχωρήσει την αποθηκευσή ενέργειας. Κατακόρυφα βλέπετε τις ε, διάφορες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, έρευνα ανάπτυξη, ολοκλήρωση αγοράς κλπ έξι συστάσεις μας είναι η έρευνα και η ανάπτυξη συμβάλλουν στη βελτίωση της ε, αλυσίδας τροφοδοσίας. Το να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην αγορά ε, για την ε, αποθήκευση του φυσικού αερίου θα βοηθήσει επίσης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανταγωνιστική αποθήκευση ενέργειας. Θα πρέπει δηλαδή να ξεφύγουμε από την την μη ευθύνη των, ε, των παραγωγών. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στις ε, αγορές. Θα πρέπει να επιτρέπεται ο έλεγχος και η ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Κλείνω διότι τελείωσε ο χρόνος μου. Θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρα Ουγκάρτε, αν έχετε και άλλες διαφάνειες να μας παρουσιάσετε. Ίσως αργότερα με αφορμή τις ερωτήσεις και τη σύντομη συζήτηση που θα έχουμε. Θα δούμε μετά τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, μπροστά σας. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Διότι για μας η άμεση ερώτηση είναι αν υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης ε, στην Ευρώπη ή όχι. Και αν ναι, σε τι βαθμό. Έβλεπα και το διάγραμμα και έβλεπα τις διαφορετικές δυνατότητες που παρουσιάζονται. Άλλο είναι τα μελλοντικά σχέδια και όνειρα και άλλο είναι, εάν τώρα ευθύ αμέσω έχουμε κάποιε λύσει, διότι μπορεί να καταλάβετε και το δικό μα πρόβλημα. Από τη μια, πρέπει να πετύχουμε του στόχου το 2020, το 2003 για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Πώ θα γίνει αυτό, εάν δεν έχουμε εναλλακτικέ. Διότι η εναλλακτική υπαριθμών 1, αυτή που τώρα έχουμε μπροστά μας, είναι να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες άντλησης, δηλαδή να αντλήσουμε νερό από λίμνες και να το αξιοποιούμε όταν δεν υπάρχει άνεμος ή ήλιος για τις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά εξ όσων κατάλαβα από την ε, παρουσίασή σας, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά άλλη εναλλακτική μπροστά μας. Και αυτή είναι και η βασική ερώτηση. Υπάρχει εναλλακτική για την αποθήκευση για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των εθνικών δικτύων και να αποφύγουμε τα blackout. Να θυμίσω ότι οι στόχοι ορίζουν 24% ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτω μέλος να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Και πολλές είναι οι χώρες που ήδη έχουν επιτύχει αυτό το 24%. Τον υποχρεωτικό στόχο του 24%. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα για τις χώρες που αισθάνονται ασφάλεια. Πίσω από τις πόρτες λένε οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 24% από ανανεώσιμες είναι επικίνδυνο και αδύνατο να ελεγχθεί λόγω των οξέων των μεγάλων, των αυξημένων τιμών της ενέργειας όταν κάποια στιγμή υπάρχει πάυση της παραγωγής λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας ή όταν δεν υπάρχει άνεμος. Υπάρχει λοιπόν κάποια εναλλακτική αυτή τη στιγμή επιτάπητος και αν ναι, ποιες είναι οι δυνατότητές μας ώστε να γνωρίζουμε, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις τεχνολογίες για τους δεσμευτικούς μας στόχους, για τις ανανεώσιμες. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή θα είναι επιβλαβής λόγω των ε, πραγματικών τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Γκροστέτ εκ Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή την ε, σύγκριση. Αλλά διερωτώ με. Βεβαίω για την ασφάλεια της ε, προμήθειας η αποθήκευση αερίου είναι καθοριστική. Αλλά και εδώ αυτό μπορεί να επιληθεί χωρίς πολλές δυσκολίες πιστεύω. Α, κατά άλλα όμως, όταν μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια, η ερώτηση που διαρκώς θέτω και την έθιξε Φευγαλέα ένας από τους προηγούμενους ομιλητές. Όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούν περαιτέρω, τι κάνουμε Ακόμη διερωτώμεθα για τη δυνατότητα που έχουμε να αποθηκεύσουμε σε μεγάλες ποσότητες την ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει διακύμανση στην παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Ε, είναι κάτι ανυπολόγιστο. Τι κάνουμε εδώ, έχουμε αρκετές επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης, έρευνας και κοινοτομίας για να δούμε βραχυπρόθεσμα τι θα γίνει, θα μπορούμε να αποθηκεύουμε με τρόπο αποτελεσματικό και ενδιαφέροντα ενέργεια προκειμένου να έχουμε περισσότερη ασφάλεια, προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και ταυτόχρονα το κόστος να μην είναι δυσβάσταχτο. Μιλώ για την τιμή των, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη στιγμή που θα μπορούμε να την υποθηκεύσουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση μου. Θα ήθελα να έχω κάποια απάντηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έριξον από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης περί αποθήκευσης. Την βρίσκω άκρως ενδιαφέρουσα αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι το εξής. Πώς μπορούμε αποτελεσματικότερα να χρησιμοποιήσουμε τη φθηνή ολική ενέργεια όταν έχουμε πλεόνασμα. Μία δυνατότητα είναι η αποθήκευση Και θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάνει κάποιον υπολογισμό. Τι θα γίνει με τις τιμές στο μέλλον, τι δείγματα έχουμε, εάν είναι δυνατόν να αποθηκεύσουμε ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των μικρών των μεγάλων όγκων αποθήκευσης, εάν θα μπορούσε αυτή να είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή για το μέλλον. Και ένας άλλος να, ε, τρόπος να υποθηκεύσουμε την ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο είναι εάν την προωθήσουμε στο σύστημα θέρμανσης και χρησιμοποιηθεί αντί αερίου. Δηλαδή να γίνει κάποια είδου αποθήκευση στο σύστημα θέρμανσης για αποτελεσματική χρήση της πολύ φτηνής όταν έχουμε το πλεόνασμα. Την έχετε κοιτάξει αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κάπελ, εκ μέρους του ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ουγκάρτε. Στην παρουσίασή σας μας δείξατε ότι η αποθήκευση ενέργειας θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να πετύχουμε την Ενεργειακή Ένωση. Και όσον αφορά την ασφάλεια της τροφοδοσίας και όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την οικονομία απειλαγμένη από άνθρακα. Είναι επίσης κάτι που θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας. Μας δείξατε ότι η αποθήκευση θα είναι μία από τις βασικές λύσεις ευελιξίας. Θα πρέπει να αυξήσουμε το δυναμικό αποθήκευσής μας και επίσης μας δείξατε πώς η, μεγάλη αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να απειλήσει την σταθερότητα της αγοράς. Γι' αυτό όσον αφορά τα ρυθμιστικά σημεία συμφόρηση. Μας είπατε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και ανάπτυξη, διότι βρισκόμαστε πίσω από τις ΗΠΑ και τη Ιαπωνία. Επίσης, χρειαζόμαστε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχετε υπολογίσει ε, τι δυναμικό χρειάζεται, αρκούν τα προγράμματα που υπάρχουν, ή θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και στο πλαίσιο του Ορίζον 2020 αλλά και σε άλλα προγράμματα που ασχολούνται με τα FEE δίκτυα. Thank you much, Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς? Δεν βλέπω να έχει κανείς άλλος ερωτήσεις. Ο κύριος Όλιβερ Κόχ είναι να αναπληρωτής επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας για την ενέργεια, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο κτλ. Ενεργειακές αγορές. Έχετε το λόγο, κύριε Κόχ. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Η το τμήμα μας μάλλον, η μονάδα μας, το τμήμα μας είναι εκείνο που ασχολείται με το τέταρτο πακέτο και με την ενεργειακή αγορά. Το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας είναι κλειδί βέβαια και για τον ε, ηλεκτρισμό και για το φυσικό αέριο. Ο σχεδιασμός για τον ηλεκτρισμό, για παράδειγμα, οδηγεί σε διάφορες ε, ιστορίες, σε διάφορα θέματα που έχουμε συζητήσει, δεδομένου ότι η, αλλάζει η ενέργεια και αντί το σύστημα ηλεκτρισμού να απορρέει από την παραγωγή, προχωράμε σε ένα σύστημα πολύ σύντομο που θα έχουμε 30, 40 και παραπάνω της 100 της ενέργειας η οποία απαιτεί αποθήκευση. Τότε δηλαδή που δεν θα έχουμε αέρα ή δεν θα έχουμε ήλιο θα πρέπει να έχουμε αποθηκεύσει ενέργεια. Οποιουσδήποτε λοιπόν σχεδιασμός νέας αγοράς είναι κάτι αναγκαίο. Και είναι πολύ καλό που υπάρχει η μελέτη με διάφορα στοιχεία μέσα. Η αποθήκευση ηλεκτρισμού αποτελεί μέρο του σχεδιασμού, όντω. Πώ δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι δεν έχουμε συνεχή ροή ενέργεια και τι σχεδιασμό απαιτείται. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και για την εμπορία ενέργεια, τι ευελιξία θα χρειάζεται μια τέτοια αγορά διασυνοριακά. Και γι' αυτό πρέπει να επιταχύνουμε ε, τα, την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Ανάλογα με το αν έχουμε άνεμο ή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Και κοιτάμε και τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την αποθήκευση. Έχουμε κάποιους κανόνες και σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και είναι πρόσδεκτο το μήνυμα της μελέτης ακούσαμε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε να αποφύγουμε την αποθήκευση και στην ομάδα για την αποθήκευση ενθαρρύνουμε και τους πολίτες, τους πελάτες ουσιαστικά να συνεισφέρουν με ιδέες στον προβληματισμό. Για να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η ζήτηση μαζί με την αποθήκευση έχουν τεράστια σημασία. Πώς ε, αν ε, αναβάλουμε την ε, αποθήκευση, την κατανάλωση της ενέργειας έστω για κάποιες ώρες, πόσο μεγάλο όφελος μπορεί να προσφέρει ακόμα και όταν αυτό γίνεται μέσα σε ένα νοικοκυριό. Κοιτάμε λοιπόν εμείς όλους του, όλα τα εμπόδια, όλες δυσκολίες που υπάρχουν και σίγουρα θα τα συζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε η αποθήκευση της ενέργειας να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του συστήματος. Ελπίζουμε ότι τεχνολογικά θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος και φυσικά θέλουμε εξέλιξη και στην ομοθεσία και όσον αφορά την κατανάλωση ε, του καθενός μας κλπ. Αυτά για τον ηλεκτρισμό. Τώρα για το φυσικό αέριο. Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Έχουμε ξεχρονίσει τις αγορές. Υπάρχει το λεγόμενο hub-based. Συμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και όσον αφορά την εμπορία. Συγχρόνως η αποθήκευση μερικές φορές είναι ε, περιττή. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τον εφοδιασμό. Όσον αφορά το χειμερινό πακέτο για το φυσικό αέριο, κάποια από τα βασικά ζητήματα που θέσατε θα ανταλάβουμε υπόψη μας. Πώς να διατηρηθεί αποθήκευση, και ποια είναι η σχέση με τον ηλεκτρισμό. Πώς δηλαδή να μοιραστεί το θέμα αυτό της αποθήκευσης στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Πώς θα χρησιμοποιηθούν διασυνοριακά επίσης τα στοιχεία αυτά. Όταν δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια είναι δύσκολα διασυνοριακά να περάσει ενέργεια. Θέλουμε λοιπόν αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό. Και κάθε περιφέρεια, κάθε χώρα, κάθε πόλη να μπορεί να αποθηκεύει τη δικιά της την ενέργεια για να μπορεί μετά να τη μοιράζεται με κάποιον άλλον σε περίπτωση που ο άλλος το χρειάζεται. Είναι πιο αποτελεσματικό να μπορούμε να μοιραζόμαστε με κάποιον άλλον την ενέργεια που έχουμε αποθηκεύσει παρά να πρέπει ο καθένας να έχει το δικό του και να λειτουργεί με αυτό. Άρα λοιπόν είναι θέμα στρατηγικής αποθήκευσης ενέργειας και σύντομα θα έχουμε να σας παρουσιάσουμε κάτι από αυτού. Ευχαριστούμε κύριος Ρόιλ. Έχω μία συμπληρωματική ερώτηση άκουσα πολλά σχετικά με την ε, σωστή και έξυπνη χρήση της ενέργειας. Ε, ακούσαμε και για την αποθήκευση του ε, φυσικού αερίου, αλλά δεν απαντήθηκε η ερώτηση πολλών συναδέρφων. Πότε μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα μπορέσουμε να αποθηκεύουμε ενέργεια με λογικό κόστος. Θα ήθελα σε αυτή την ερώτηση απάντηση, δεν έχω ακούσει όμως ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Το ίδιο ακριβώ θέλω να ρωτήσω κι εγώ. Όταν ε, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με περισσότερη ευθύνη ο κάθε πολίτης και ότι πρέπει να συμμετέχουν στην αποθήκευση και οι πολίτες και τη... να βοηθούν τη βιομηχανία κτλ. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό μου φαίνονται ευσεβείς πόθη. Μα το μόνο πρόβλημα είναι η αποθήκευση του ηλεκτρισμού. Όταν θα μπορούμε με μεγάλο όγκο να αποθηκεύουμε τον ηλεκτρισμό, τελείωσε, το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ειλικρινά δεν ε, ακούω λύσει. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρτέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει παραγωγή καθαρής ενέργειας και μπορεί να αποθηκευτεί. Είναι ο ηλεκτρισμός από την ε, υδρολική ενέργεια. Ξέρω ότι δεν είναι αυτή η συζήτηση ακριβώς, αλλά μερικές χώρες υποχρώνονται να ανοίξουν την αγορά τους και η δικιά μου θα αναγκαστεί να αποχωριστεί κάποιες επιχειρήσεις ε, τέτοιες ενέργειας. Κι όμως σε μερικές ε, περιοχές της Γαλλίας, στα Πυρηναία για παράδειγμα, η δραστηριότητα ε, τροφοδοτείται έτσι. Και αν δεν έχουμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις μεθαύριο, να ξέρετε ότι δεν θα έχουμε αρκετή απόδοση. Η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που είναι η τροφοδότηση με ενέργεια ολόκληρης της επικράτειας, είτε ιδιωτική, είτε ατομική, είτε συλλογική. Οπότε δεν καταλαβαίνω τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή, εν πάση περιπτώσει, όπω την καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι προ το γενικό συμφέρον. Πρόεδρος, ναι, είμαστε σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο τρίτος είναι πολύ. Δεν έχουμε χρόνο. Εσείς ήσασταν στον πρώτο γύρο μου, σωστά, οπότε ακούω την ερώτησή σας. για τις ιδιωτικές εταιρείες. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ποιο είναι το συμφέρον των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωραία. Θα σας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για να τελειώσουμε τον πρώτο και δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Μετά έχουμε απαντήσει από την Επιτροπή και από τον ομιλητή μας. Έχουμε δύο θέματα. Την αποθήκευση φυσικού αερίου και την αποθήκευση ηλεκτρισμού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από πλευράς αποθήκευση φυσικού αερίου θα μπορούσαμε να είχαμε ρυθμιστικά προβλήματα, πλησίωση, ιδιοκτησία. Και θα έπρεπε να απαντηθούν πολύ συγκεκριμένα. Αλλά ο ηλεκτρισμός είναι τελείως διαφορετικό, όπως είπανε και οι συνάδελφοι. Έχουμε βέβαια τη δυνατότητα ε, να έχουμε μια ισορροπία στα δίκτυα. Γίνεται. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα βελτιώσουμε την έρευνα γιατί ήταν κάτι που είπανε πολλοί από εσά. Ίσως θα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα από το Horizon 2020. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για διαγωνισμούς. Οπότε, αν μπορείτε να μας απαντήσετε χωριστά για το φυσικό αέριο και χωριστά για τον ηλεκτρισμό και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την έρευνα κυρίως στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Ωραία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και θα ακούσουμε τις απαντήσεις της Επιτροπής και του ομιλητή μας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να αποπειραθώ. Είναι δύσκολη ερώτηση να με ρωτάτε πότε η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι πανέτοιμη. Η απάντηση είναι δίτυχη. Εξαρτάται από το σύστημα Όπως είπε ο Γερμανός ε, συνάδελφος, έχουμε πάμπολους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία ήδη και ε, ο αριθμός διαρκώς αυξάνεται. Η ισοτιμία του δικτύου στη σελίδα 51, κοιτάξτε τη μελέτη, εννοεί ότι οι μικροί παραγωγοί από ηλιακή ενέργεια ήδη έχουν καλύτερες λύσεις να προσφέρουν. και δεν χρειάζονται τεράστιες επιδοτήσεις για να έχουν επικερδή παραγωγή. Τα έχουν καταφέρει ήδη, δηλαδή αυτή η εναλλακτική έχει ήδη φέρει καλές λύσεις. Τώρα στη Γαλλία με ε, κάποια κορύφωση στο κρύο και τεράστιες ποσότητες ενέργειας απα... απαραίτητες για την ε, θέρμανση, ε, σίγουρα η πυρηνική ενέργεια είναι η πρώτη λύση, αλλά θα μπορούσαμε τα κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης να τα αξιοποιήσουμε για να πείσουμε για την τεράστια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ότι είναι προτιμότερη η κάλυψη όταν υπάρχουν διαλύσεις στο σύστημα με τεχνολογικές βελτιώσεις ή οποιασδήποτε τεχνολογίες αποθήκευσης. Βέβαια πέραν αυτού μπορεί να είμαστε εδώ ότι οι ιδιωτικές εταιρείες, η Τέσλα και πολλές άλλες που αναφέρονται στην έκθεση ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Οπότε ναι, ε, σαφώς στηρίζουμε την έκκληση για χρηματοδότηση στον τομέα. Είναι από τους πιο ευθύς τρόπους να ταπανίσουμε τα διαθέσιμα ποσά, διότι η υποστεθέμενη αξία θα είναι τεραστία. Η δεύτερη ερώτηση, εάν καλά κατάλαβα, ήταν πώ μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει ασφάλεια στην προμήθεια από ιδιωτικέ εταιρείε, εφόσον αυτέ αναλάβουν, ε, με περισσότερα εμπορικά συμφέροντα και αν θα υπάρξει ενδεχομένω κίνδυνο λόγω της πολιτικής που θα στραφεί προς την αγορά και ίσως σε απόκεντρες περιοχές να κινδυνεύσει η ασφάλεια στην ε, προμήθεια, εάν ε, βασιστούμε στις ανάγκες της αγοράς. Το ε, διερευνούμε πολύ σοβαρά. Ουδέποτε θα επιτρέπαμε στην νομοθεσία να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αφήσουν την παραγωγή σε κάποιες περιοχές και νομίζω αυτό το έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Πέραν αυτού βεβαίω, αυτό που χρειαζόμαστε και πρέπει να το τονίσω, γιατί είναι το βασικό μας δίδαγμα από την κρίση του αερίου, είναι κάτι από αυτό που τώρα βλέπουμε να συμβαίνει και με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, δεν είναι η ιδιωτικοποίηση απαραίτητο που πλήττει την ε, ασφάλεια στην παροχή, αλλά ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση, αρκετός ανταγωνισμός, αρκετή ολοκλήρωση της αγοράς με ε, τους γείτονες. Οπότε ανεβαίνει και το κόστος της ενεργειακής παροχής. Άρα η ολοκληρωμένη αγορά παραμένει μια από τις ε, βασικότερες απαντήσεις για να είμαστε βέβαιοι για την ασφάλεια στην παροχή. Το αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ασφάλεια της παροχής. Η νομοθεσία είναι προτιμότερη λύση. Είναι μια λύση πιο επιτυχής. Και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει σε επίπεδο χώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίες κουβέντες και ανακεφαλαίωση της συζήτησή μας από τον ε, κύριο ομιλητή μας. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις σας, αυτό ακριβώς αποδεικνύουν. Το πρόβλημα είναι περίπλοκο. Από τη μια και για το αέριο και για την ηλεκτρική ενέργεια. Ή να πάω ένα βήμα ακόμη παραπίσω. Για το αέριο, τον ηλεκτρισμό, για την αποθήκευση. Ένα είναι το κόστος και από την άλλη η οργάνωση της αγοράς. Το κόστος της λύσης είναι ένα πρόβλημα που ε, αυτοεπιλύεται λόγω του δυναμικού χαρακτήρα του χώρου του ίδιου. Διαρκώς υπάρχει βελτίωση, οι διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις Το ότι μπορεί να έχουμε ανταγωνιστική τιμή είναι κάτι που ρίχνει το κόστος. Σε κάποια στιγμή θα είναι ανταγωνιστικά αυτά που θα ισχύσουν. Πότε ακριβώς δεν είναι γνωστό. Μια ερώτηση ήταν πότε λοιπόν ε, για τους τελικούς χρήστες ίσως του χρόνου. Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκού πάνελ στη Γερμανία με μια συσκευή για αποθήκευση θα αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστική προς την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου του χρόνου. Όχι σε 5 και 10 χρόνια, του χρόνου κιόλα. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάξουμε την περίπτωση της Γερμανίας που δεν έχει τόση ηλιοφανία. Εγώ έχω το παράδειγμα της Καταλωνίας από που είμαι. Αλλά δείτε και τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί υπάρχει ταχεία πρόοδος. Η διοργάνωση της αγοράς ε, παρουσιάζει ιδιαίτερα περίπλοκα προβλήματα, διότι όταν διοργανώνει κανείς την αγορά, όλο και κάτι κερδίζει και όλο και κάτι ε, χάνει. Οπότε πρέπει να κανείς πολύ προσεκτικός, με πολλή σκέψη, μελέτη και πολύ συζήτηση. Ο πρόεδρος μου ζήτησε να ξεχωρίσω τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια και το αέριο. Ναι, γιατί το επίπεδο των λύσεων είναι διαφορετικό και είναι και δύο διαφορετικά ζητήματα. Το αέριο για τους χρήστες, ηλεκτρισμού, θέρμανσης κλπ. Το αέριο λοιπόν στην Ευρώπη προς την αποθήκευση δεν είναι πρόβλημα συνολικά. Έχουμε αρκετή αποθήκευση αερίου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η αγορά δεν λειτουργεί εύρυθμα σε ορισμένες περιοχές. Συγκεκριμένε περιφέρειες. Συγκεκριμένα στις χώρες της Βαλτικής, τη Βουλγαρία, περιοχές που είναι περισσότερα απειλούμενες αν υπάρξει κάποια έλλειψη, κάποιο έλλειμμα αερίου. Και το πρόβλημα δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο, ε, δεν απαιτεί επενδύσει, απλώ χρειάζεται καλύτερη διοργάνωση τη αγορά. Η λύση ήδη παρουσιάστηκε από την Γενική Διεθνή Ενέργεια. Είναι η κατανομή, μοίρασμα. Δηλαδή, θα έχω πρόσβαση στην αποθηκευμένη ενέργεια τη χώρα γείτονο και θα έχουν πρόσβαση στη δική μου ε, αντιστροφή των ροών. Αυτό επιτρέπει την αμοιβαία κερδοφορία κάποιο που να κερδίζει από όλο αυτό. Οπότε να είναι σαφέ ε, και εύκολο για όλου είναι ο στόχο. Και επίση πάντοτε να θυμόμαστε, για να απαντήσω και στη δική σα ερώτηση, η αποθήκευση δεν θα λύσει τα προβλήματα ελλημάτων αερίου. Η αποθήκευση απλώ μετατοπίζει το πρόβλημα. Είναι ένα μαξιλαράκι σε φάση αναμονή μέχρι να πάρει κανεί το αέριό του. Δεν παράγει από μόνη τη αποθήκευση αέριο. Δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας, πέραν του να καθιστά την αγορά αποτελεσματικότερη και να υπάρχει καλύτερη κατανομή σε επίπεδο ένωσης κιόλα. Θα πρέπει ούτω ή άλλω να διαφοροποιηθούν οι πηγέ παροχή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αποθήκευση αερίου, τι πρέπει να γίνει. Να ξαναδεί κανεί την ποσότητα αερίου που ε, καταναλώνεται, διότι έτσι κι έξω θα έρθει από κάπου. Και δεύτερον, διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση των οδών παροχή. Αυτά για το αέριο. Για τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός είναι μια διαφορετική περίπτωση, διότι οι τεχνολογικές λύσεις είναι σε πολύ διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Κάποιες λύσεις είναι πολύ ε, ανταγωνιστικές, όπως η άντληση αποθήκευση μεσοάντλησης. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ένα υψόμετρο, μπορεί κανείς να πάρει το νερό, να το αντλήσει, να το πάει εκεί και να αποθηκευθεί ε, ε, αέριο. Να σας ξαναπάω στην παρουσίαση. Μπορούμε να ξαναδούμε την διαφάνεια. Έχετε ξεπεράσει τα 5 λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Αυτή είναι μία λύση, μία λύση που ήδη είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Η άλλη ορίζει ότι σε άλλο επίπεδο της κλίμακας, σε άλλο ύψος της κλίμακας, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από το τελικού χρήστη, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι πολύ μικρές ποσότητες εκεί. Αλλά τι θα γίνει αν είναι πολλοί, όπως η Γερμανία, λόγω χάρη, πολλοί έχουν τέτοιες συσκευές. Κάτι που αναμένεται να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, το έχει αναλάβει η Τέσλα. Τόσες μπαταρίες περιμένουμε του χρόνου. Δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η λύση. Δεν συνηγορώ υπέρ αυτής της λύσης, απλώς είναι πράγματα που συμβαίνουν. Ήδη ε, λαμβάνουν χώρα, όπως τα κινητά μας έχουν πλέον καλύτερες μπαταρίες που κρατάνε περισσότερο. Είναι λύσεις που έρχονται, συμβαίνουν ήδη. Αυτό δείχνει ότι η λύση δεν είναι κάτι το θεωρητικό όπως το φανταζόμασταν πριν από 30 χρόνια που θα υπήρχε μια μεγάλη λύση για να λυθούν όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα. Και πριν τέσσερα χρόνια φανταζόμασταν ότι μία λύση κεφαλαιώδης θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όχι, έχουν αλλάξει οι λύσεις, το είδος των λύσεων και το είδος των προβλημάτων. Και εμείς, και εμείς οι χρήστες, οι καταναλωτές, είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι, μετακινούμαστε. Η λύση δεν θα είναι μία και μία, θα είναι ένας συνδυασμός λύσεων. Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία από τις λύσεις δεν θα είναι η μία και μόνη. Ένα, δύο... Ηλεκτροκινητικότητα. Δεν πρόλαβα να το αναπτύξω, αλλά δείτε τα μεγέθη, τις τάξεις μεγεθών στην διαφάνεια αυτή. Δείχνει το διάγραμμα τη δυνατότητα αποθήκευσης από, τις, ε, από τους πόρους υδροάντλησης το 2014. Αυτό είχαμε πέρσι στην Ευρώπη και την ερχόμενη εβδομάδα κάτι που δεν φαίνεται, είναι μικροσκοπικό εκεί για το 2014, είναι ο όγκος ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύτηκε από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα τα πάρκινγκ, σε στάθμευση, ε, είναι ούτως ή άλλως συνδεδεμένα με το δίκτυο αυτά. Δεν φαίνεται καν στο διάγραμμα, αλλά υπάρχει. Οι υπολογισμοί μας, δείτε το σκούρο μπλε, λένε ότι το στο 2030 με 14% περισσότερα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην αγορά θα έχουμε το σκούρο μπλε κομμάτι, δυνατότητα αποθήκευσης και συνδεδεμένο με το δίκτυο σε σύγκριση με το γαλάζιο, την ε, υδροάντληση και δείτε τι γίνεται με αυτό το σενάριο που είναι και επιφυλακτικό εφόσον έχουμε ηλεκτροκινητά οχήματα, περισσότερα ηλεκτροκινητά ε, οχήματα στην αγορά. Βεβαίω και αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην αγορά, θα συνεχίσουν να μπαίνουν, αλλά δεν οδηγούμε στο κινητό διαρκώ. Τι περισσότερε στιγμέ είναι σταθμευμένα τα οχήματα και είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. Η νομοθεσία και η διοργάνωση της αγοράς θα αξιοποιήσουν ή όχι αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια. Αυτό είναι μια ερώτηση που έρχεται έπειτα. Αλλά δεν απαντώ σε αυτό τώρα. Απαντώ μόνον στο πότε. είναι ε, θέμα των πολιτικών ηθινόντων και σχεδιασμού πολιτικής να αποφασίσει εάν η αγορά θα διοργανωθεί έτσι ή αλλιώς. Γιατί πάντοτε υπάρχουν ε, κέρδη και απώλειες. Με ποιο τρόπο, σε τι επίπεδο, λιγότερο ή περισσότερο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω, να το απαντήσω εγώ. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Έχω την άποψή μου, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν η αποθήκευση είναι μία από τις πολλές λύσεις. Αλλά και η ίδια η αποθήκευση, η αποθήκευση αυτή καθεαυτή δίνει μια πλειάδα δυνατοτήτων που δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουμε σε λίγα λεπτά. Η ε, αποθήκευση θέρμανσης. Όντως η Ευρώπη προηγείται εδώ. Προηγείται και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας και της Κορέας και της Κίνας. Η αποθήκευση θέρμανσης για τη χρήση και για τη μετατόπιση αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ πετυχημένη. Και δεν είναι για κάποια τεχνολογία φοβερά προηγμένη. Είναι προγράμματα που ήδη υπάρχουν στο, στα πλαίσια του 2020. Τώρα, πόσο περισσότερο θέλουμε από τις επενδύσεις του 2020, ίσως το διπλάσιο από αυτό που τώρα επενδύεται το διπλάσιο από το ποσό που προβλέπεται για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο. Να θυμόμαστε ότι όπως τα κινητά μας που αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερες μπαταρίες και τα αγοράζουμε έτσι κι αλλιώς, τα αγοράζουμε από κάποιον που τα παράγει ίσως στην Κορέα στο μέλλον. Αναλόγως θα αγοράζουμε τις συσκευές μας που θα κάνουν και αποθήκευση ενέργειας από τους αυτούς μας ίσως, αλλά ίσως από κάπου αλλού. Εκεί είναι το ερώτημα. Και είναι μέρος ε, της όλης μας ε, έρευνας. Αυτά, Πρόεδρε. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα για να μπορέσω να απαντήσω. Ένα λεπτό μπορείτε. Σας φτάνει. Ένα λεπτό σας το δίνουμε. Εντάξει. Δύο. Δύο λεπτά. Οπότε, θα σας ενθάρρυνα για τα θέματα τα τεχνικά που είναι τόσο ποικίλα και για τα θέματα του κόστους να δείτε την έκθεση αυτή που είναι αρκετά εκλεκευμένη. Ε, δεν απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες της ενέργειας, απευθύνεται σε ηθήνοντες πολιτικούς, αυτούς που σχεδιάζουν και λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις με γενικές ερωτήσεις. Πόσο κοστίζει, πόσο αξία έχει το ένα ή το άλλο. Και έπειτα, εάν μπορούσα να συνεισφέρω εγώ στον ε, ε μιλήσω στο κοινοβούλιο, το ευρωκοινοβούλιο, κάτι που με ενδιαφέρει είναι πώς θα διοργανωθούν καλύτερα οι αγορές. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνετε, είναι πρόσδεκτη. 20 δευτερόλεπτα. Έχω μπερδευτεί πιο πολύ από ό,τι πριν από δύο λεπτά. Ε, ο Επίτροπος Καλνιέτη ήρθε πριν από λίγους μήνες και μα είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη ε, κλίμακας διάδοση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διότι δεν υπάρχει δίκτυο. Και μα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαμε να έχουμε πάνω από 10 ηλεκτροκίνητα ανά δρόμο. Αυτή ήταν η δήλωση του Επιτρόπου Καλνιέτε προσφάτω. Τώρα εσείς έρχεστε και μας λέτε ότι η στρατηγική είναι να βασιστούμε στο μεγάλο αριθμό ηλεκτροκινήτων οχημάτων και θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης ως εξ επιτούτου. Δεν καταλαβαίνω τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχουν τα ηλεκτροκινήτα οχήματα ή όχι. Θα βασιστούμε στα στρατηγική μας τα ηλεκτροκινήτα οχήματα ή όχι. Και ακόμα ένα σχόλιο. Είστε λέτε σοβαρά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στρατηγική, δυστυχώ δεν ακούει ο πρόσωπό τη γιατί μόλι έφυγε, που λέει ότι σε ένα εργοστάσιο θα ζητάμε από του εργάτε να έρχονται στι 8 και θα λένε ότι στι 11 λόγω τη τιμή τη ενέργεια θα σταματάμε, θα κάνουμε μια διακοπή και μετά θα ξαναρχίζει η παραγωγή στο εργοστάσιο. Και επιπλέον, οι καταναλωτές από 9 ως 1 που είναι ξύπνοι, τι θα κάνουν σπίτι τους. Πώς θα ανοιγοκλίνει κανείς τις συσκευές μετά από τέτοια μακροσκελή ομιλία δεν θα υπάρξει απάντηση. Την επόμενη φορά στην επόμενη συνεδρίασή μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν ε, πολύ μακρά η όλη μας συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις και ευχαριστώ και εσάς ε, συνάδελφοι για την ε, θερμή σας συμμετοχή. Νομίζω ότι ήδη είχαμε κάποιε πρώτε ικανοποιητικέ απαντήσει. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Ουγκάρτε, και για την παρουσία σα και για την μελέτη σα για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Αποθήκευση τη ενέργεια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ εγώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να σα βοήθησα. Ωραία. Επόμενο σημείο. Άσυρ, έκθεση παρακολούθηση τη αγορά και άλλες ενεξελίξει δραστηριότητε. Παρουσιάσεις από δύο εκπροσώπους της ΆΣΕΡ, της Ένωσης ε, του Φορέα για τη Συνεργασία των Ρυθμιστών Ενέργειας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διευθυντής της ΆΣΕΡ. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε. Συναντιόμαστε από καιρού εις καιρών. Είναι σημαντικό για μας στην, έκθεση για την, στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της αγοράς. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή. Και να θυμίσω σε όλους σας ότι είναι το, η τρίτη δεσμή για την ενέργεια που ζητά από τον οργανισμό την Άσερ να διοργανώσει την συνεργασία των ρυθμιστών ενέργειας και να παρακολουθήσει την αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο. Η τελευταία εκδοχή της ε, έκθεσης δημοσιεύτηκε σήμερα κιόλας, 30 Νοεμβρίου. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας παρουσιάσετε την έκθεση. Έχετε την επιλογή ποιος θα ξεκινήσει. ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο διευθυντής της Άσερ, του Άσερ μάλλον. Έχετε την επιλογή. Ο Λόρντ Μόγκ. Δεν χρειάζεστε συστάσεις, διότι έχουμε συναντηθεί επανειλημμένος ε, στη συνεδρία της Επιτροπής Ήτρε. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομο, θα χαρείτε που θα το ακούσετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Σήμερα το μεσημέρι εκδόθηκε η έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τη βοήθειά της ε, στο, όσον αφορά τους πόρους το Κοινοβούλιο επανειλημμένα ε, μας προσέφερε πολύτιμη βοήθεια και νομίζω το 2016 ακόμα περισσότερο. Σκοπός ε, αυτής της παρουσίασης είναι να σας παρουσιάσουμε τα βασικά ε, στοιχεία με βάση τα δεδομένα που συλλέξαν το 2014. Τα συλλέξαμε λίγο νωρίτερα από την πέρσι, αλλά υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να μπορέσουν να συντάξουν τα στοιχεία. 387 σελίδες ε, μπορείτε να κάνετε να διαβάσετε απόψε και αύριο. Μπορούμε να σας κάνουμε και τεστ μετά αν θέλετε. Ε, σας έχουμε δώσει όμως και μία σύνοψη και διαφάνειες σε περίπτωση που κάποιος από τους συναδέλφους σας, το προσωπικό σας ε, θέλει να εξετάσει την έκθεση. Ο λόγος που έχουμε μια τόσο αναλυτική έκθεση είναι ότι νομίζουμε ότι έτσι θα έχουμε βαθύτερη ανάλυση των ε, μελλοντικών θεμάτων που θα προκύψουν του χρόνου. Θα ήθελα να τονίσω τον κεντρικό ρόλο του καταναλωτή. Κοιτάμε το θέμα από πλευράς του καταναλωτή. Να προχωρήσω λοιπόν τώρα στα στοιχεία της έκθεσης. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα θέλαμε να αναφέρουμε. Δεν θα πω όμως σε πολλές λεπτομέρειες. Όσον αφορά την υποχρέωση παροχής σε δημοσίων υπηρεσιών, ε, έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, αποσυνδέσεις δεν παρακολουθούνται παντού, αλλά σε πολλές χώρες και έτσι έχουμε αρκετές χρήσιμες πληροφορίες. Θα ήθελα να αναφερθώ πιο αναλυτικά στους ευάλωτους καταναλωτές, διότι νομίζω ότι οι συνάδελφοί σας ε, θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Όσον αφορά την πληροφόρηση προς τους καταναλωτές, βλέπουμε διαφορετική εφαρμογή των κανονισμών και πολύ συχνά εχθρός του καλού ε, είναι το καλύτερο. Τα, οι ευφυείς ε, μετρητές ε, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, όχι όμως παντού και κατόπιν θα περάσουμε στα παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν κάποιες διαφάνειες. Καταρχάς όσον αφορά τον ευάλωτο καταναλωτή υπάρχει υποχρέωση του να έχει κανείς ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή, ο ορισμός αυτός όμως ποικίλει από χώρα σε χώρα. Έχουμε ρητούς ορισμούς και άλλους ε, που εννοούνται. Περίπου τα μισά κράτη-μέλη έχουν τέτοιον ορισμό ε, και θα δείτε για παράδειγμα τις διαφορές ανάμεσα στη Βουλγαρία, τη Φιλανδία και, και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, στα παραδείγματα που σας δίνουμε. Όσον αφορά τους ευφυείς μετρητές, βλέπετε στις κίτρινες χώρες στο τέλος του 2014 λιγότερο από το 10% των οικοκυριών είχαν ευφυείς μετρητές και υπάρχουν και άλλες χώρες όπου είναι πολύ υπαλλοί μετρητές. Βλέπετε ότι το μισό των ε, κρατών μελών ήδη έχουν ε, εφαρμόσει τις ελάχιστες ε, τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις στην νομοθεσία τους. Κατόπιν, περνώ στα παράπονα των καταναλωτών. Βλέπετε το πράσινο δείχνει τα παράπονα που έχουν να κάνουν με την τιμή και την έκδοση των λογαριασμών. Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ενδυνάμωση του καταναλωτή, σε κάποιε δικαιοδοσίε ε, θα πρέπει να οριστεί ο ίστατος προμηθευτή ε, και όσον αφορά το φυσικό αέριο και όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί μια, ένα ελάχιστο τεχνικών λειτουργιών για τους ε, ευφυείς ε, μετρητές ε, και τέλος χρειάζεται παρακολούθηση σε αρκετούς τομείς διότι αυτή τη στιγμή γίνεται ανεπαρκής παρακολούθηση σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα είναι η διακοπή του ρεύματος επειδή δεν έχει πληρωθεί ο λογαριασμός κλπ. Και δίνω το λόγο στο συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ ε, σαφείς παρατηρήσεις σας ε, τώρα στην αρχή της συζήτησής μας. Ο κύριος Ποτόσνικ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για την στήριξή σας στην, στον οργανισμό μας. Τα αποτελέσματά μας είναι θετικά, ίσως όχι τόσο θετικά όσο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα είναι θετικά. Τι θα καλύψω λοιπόν εγώ τώρα, τις λιανικές αγορές πρώτα απ' όλα. Και πριν αρχίσω να σας παρουσιάζω κάποια αποτελέσματα, να σας πω ότι κανονικά είναι πιο μεγάλη η έκθεσή μας και μόνο παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάτι το οποίο είναι προφανές για όλους, ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει και που κάνουμε τα τελευταία χρόνια για να προωθήσουμε μια ελεύθερη αγορά, πρέπει να είναι προς του καταναλωτή. Οπότε το κέντρο για μας είναι ο καταναλωτής. Τα ωφέλη είναι για τον καταναλωτή. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Για να δούμε λοιπόν σε τι βαθμό έχουμε βοηθήσει τους καταναλωτές. Ας δούμε πρώτα τη χοντρική αγορά. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε δύο τάσεις. Από τη μια μεριά η ζήτηση πέφτει. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και το 2014. Όλα τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ είναι το 2014 παρεμπιπτόντως. Και άλλη τάση είναι η αύξηση των ανανεώσιμων για να ε, φτάσουμε το στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα είναι μείωση των τιμών χοντρικής, χοντρικής συνολικά, κάτι το οποίο δεν εκπλήσει κανένα. Αν δούμε στους κόμβους, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν πέσει γύρω στο 50 με 80%. Είναι αξιοσημείωτη η μείωση δηλαδή των τιμών. Η άλλη πτυχή τώρα είναι ότι προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τις αγορές. Έχουμε ένα σχέδιο για να βελτιώσουμε την ικανότητα διασύνδεσης, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι την ικανότητα που ήδη διαθέτουμε πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε πλήρως και πιο αποτελεσματικά. Δύο διαφάνειες έχω εδώ. Η μία δείχνει τι ικανότητα διαθέτουμε για διασυνοριακό εμπόριο. Ποιο είναι το ποσοστό της αγοράς δηλαδή. Ολόκληρο το κατάλογο τον έχετε στην έκθεση. Εδώ έχουμε την Αυστρία προς τη Τσεχία, από Γερμανία προς Γαλλία, από Ελβετία προς Γερμανία και από Γερμανία προς Πολωνία. Και η σύγκριση εδώ είναι, είπαμε, της ικανότητα. Δεν λέμε ότι πρέπει να είναι πλήρης, αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι η ικανότητα για να είναι μόνο ένα μικρό μόνο ποσοστό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να διθέσουμε περισσότερη ικανότητα και αν δούμε ανάμεσα στην Γερμανία και την Πολωνία βλέπετε ότι λείπει μία, μία στήλη. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να υπάρξει σύνδεση τη αγορά στην Ευρώπη και την απο... πώ αποτελεσματικά χρησιμοποιεί το... η δυνατότητα που προβλέπετε το 2014 στο 86% των περιπτώσεων στην Ευρώπη εξοποιηθηκαν αυτές οι δυνατότητες στη σωστή κατεύθυνση. Στις προηγούμενες παρουσιάσεις τις περασμένες χρονιές έλεγα ότι κάποιες δυνατότητες διασύνδεσης έστειλαν την ενέργεια σε λάθος κατεύθυνση. Νομίζω ότι με την σωστή διασύνδεση της αγοράς αυτό αποφεύγεται και είναι ένα θετικό σημείο. Το τρίτο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ είναι για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας οι μηχανισμοί δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται. Δεν θα είναι έκπληξη για εσάς γιατί σα απασχολεί εδώ και χρόνια ότι μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων είναι ε, κάποιοι μηχανισμοί που έχουν ήδη εισαχθεί και κάποιοι που μελετώνται. Αυτό που μας απασχολεί είναι όχι απλώς οι μηχανισμοί και το κατά πόσον μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά ότι εφόσον δεν υπάρχει συντονισμό μπορεί να στραπλαθεί η εσωτερική αγορά. Ποιε είναι λοιπόν οι συστάσει μα. Όσον αφορά την αγορά ενέργειας. Στην έκθεση βέβαια θα διαβάσετε πολύ περισσότερο. Το πρώτο είναι ότι προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την ε, ικανότητα διασύνδεσης εμπορικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίσουμε εκ νέου και πιο συντονισμένα την ικανότητα που μπορεί να διατεθεί σε διάφορα πλαίσια αγοράς. Πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα γίνουν οι υπολογισμοί και να διασφαλίσουμε στη συνέχεια ότι διασυνοριακά οι ανταλλαγές και μέσα σε μια ίδια δικαιοδοσία θα αντιμετωπίσονται με τον ίδιο τρόπο. Ισότιμα, κάτι το οποίο δεν ισχύει τώρα. πρέπει να υπολογίσουμε καλύτερα την ε, διαθέσιμη ικανότητα. Και έπειτα πρέπει να καλύψουμε και τις περιοχές που δεν καλύπτονται και να διασφαλίσουμε ότι πρώτα τα αρμότι φραγμούς υπάρχουν στο θέμα του εμπορίου, πέρα από την ικανότητα που είπαμε ότι πρέπει να υπολογίσουμε την ασφάλεια, την σωστή αξιολόγηση, και αν θέλουμε έναν μηχανισμό ικανότητας να τον σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην στρεβλώνεται το εμπόριο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα στον αφορά το φυσικό αέριο. Εδώ βλέπουμε μια θετική τάση. Με τους κόμβους να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι τιμές έχουν πέσει το 2014. Βλέπουμε επίσης εδώ και τη σύγκληση τιμών ανάμεσα σε κόμβους και ανάμεσα σε κόμβο και μακροχρόνια διμερές εμπόριο. Βλέπω ότι οι αγορές γίνονται πιο ολοκληρωμένες. Αν δούμε τις τιμές είναι και το κόστος, είναι σημαντικό να δούμε ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορές ανάλογα με την περιοχή. Έχουμε το TTF στις κάτω για παράδειγμα, και εδώ φαίνεται η διαφορά στις χώρες μέλη και στο TTF. Και το συμπέρασμα είναι το κίτρινο κομμάτι δεν υπάρχει διαφορά, στο ανοιχτό μπλε υπάρχει μια μικρή διαφορά και στο μπλε σκούρο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την εγκύτητα όσο με τη ρευστότητα της αγοράς. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μεγαλύτερη σημασία στην βελτίωση της ρευστότητα των hubs φυσικού αερίου. Για κάποια ευαίσθητα σύνορα παίζει ρόλο η ρευστότητα, πολύ μεγάλο. Όταν δεν υπάρχει η αντιστροφή της ροής. Ποια είναι τα συμπεράσματα. Πρέπει να έρθουν οι φραγμοί, τα εμπόδια όσον αφορά τους κόμβους, να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα, να υπάρχει εμπόριο hub to hub και προμήθεια έτσι ώστε να διευκολύνονται οι τιμές. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε τις επενδύσεις και να ολοκληρώσουμε τους κόμβους και τις αγορές προκειμένου να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή διασυνοριακή αγορά. Τώρα όλα αυτά πώς επηρεάζουν τον καταναλωτή. Εδώ έχουμε το πρώτο θετικό στοιχείο. Είναι τουλάχιστον για τους καταναλωτές ενέργειας βλέπουμε να αντιστρέφεται η τάση σε σχέση με παλιότερα και να μειώνονται οι τιμές. Για τα νοικοκυριά όμως δεν ισχύει αυτό ακόμα. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά λοιπόν στη τάση. Το στοιχείο ενέργεια στις λιανικές ε, τιμές αλλάζει η συμπεριφορά ανάλογα με τις χώρες. Εδώ βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις χωρών Αυστρία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπουμε ότι για τη βιομηχανική κατανάλωση υπάρχει ε, πιο μικρή διαφορά ανάμεσα στη τιμή χοντρικής και λιανικής. Ενώ όταν πρόκειται για τα νοικοκυριά υπάρχει απόκληση. Γιατί. Πρώτον, γιατί υπάρχει περιορισμός της αρμοδιότητας ανάμεσα με τις αγορές. Και ο ανταγωνισμός περιορίζεται, είναι το κομμάτι το μπλε που βλέπετε, το σκούρο. Ενώ στον ηλεκτρισμό πέφτει στο 40% το 2014, που είναι τέλη με αφιζητούσιμα. Αυτή είναι η μία πτυχή η άλλη είναι το θέμα της επιλογής του καταναλωτή. Έχει μία ευρή επιλογή. Υπάρχουν διάφορες προσφορές για τον καταναλωτή, κάτι το οποίο δείχνει οριμότητα. Εδώ είναι οι εθνικές αγορές σε κατηγορίε ανάλογα με το πότε υπήρξε η ελευθέρωση, λιγότερο από 5 χρόνια πριν, 5 με 10 χρόνια πριν ή πάνω από 10 χρόνια και βλέπετε τον αριθμό των διαφορετικών επιλογών που έχει ο καταναλωτή που είναι όλο και περισσότερε. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Τέλο, τελευταία μου διαφάνεια. Είναι κάτι που κάθε χρόνο παρουσιάζουμε και το βρίσκω πολύ καλό, γιατί πρόκειται για μια σύγκριση. Να δούμε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην εξοικονόμηση που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά. Παλιότερα λέγαμε ότι είναι πρόβλημα. Τώρα δεν είναι τόσο. Γιατί οι καταναλωτές δεν προσελκύονται μόνο από τις χαμηλές τιμές, αλλά και από άλλα στοιχεία. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τη διάκριση, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που εμποδίζει τον καταναλωτή να αλλάξει προμηθευτή και τι όχι. Να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά, συνεπώς, όλων των προσφορών. Τέλος φέτος για πρώτη φορά η... σιγάγαμε, και έναν ε, δείκτη για τα επίπεδα ανταγωνισμού και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η θέση στις διάφορες αγορές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην έκθεση, αλλά εδώ βλέπετε τις χώρες όπου τα πάνε καλύτερα όσον αφορά τον ηλεκτρισμό ή το φυσικό αέριο. Για τον ηλεκτρισμό είναι οι βόρειες χώρες πιο πολύ, για το φυσικό αέριο οι άλλες που βλέπετε τη διαφάνεια. Τελικά, οι συστάσεις μας για να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις είναι να προωθήσουμε την είσοδο στην αγορά, άροντας τα εμπόδια, να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται τι αγορές καλύτερα. Χρειάζονται πληροφορίες και χρειάζεται να πάψει να υπάρχει προκατάληψη κατά της αλλαγής προμηθευτή να διευκολύνουμε δηλαδή τον καταναλωτή στην οτροπία της αλλαγής. Αυτά είναι τα κύρια. Και συγγνώμη αν σε 10 λεπτά χρειάστηκε να σας διηγηθώ τόσες σελίδες. 14 λεπτά ακριβώς, ναι. 14 λεπτό είχαμε στα 8, στα 10 λεπτά και το είπατε και στα 14 λεπτά. Τρεις φορές είπατε τελικές παρατηρήσεις. Δεν ήθελα όμω να σα σταματήσω γιατί όλα ήταν τελικέ παρατηρήσει. Τέλο πάντων, πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσει. Σα ευχαριστώ και του δύο για τι φοβερέ σα ομιλίε, ω συνήθω. Και να ζητήσω από του συναδέλφου να πάρουν το λόγο. Η κυρία Κάλλα, η κυρία Κάπελ, ποιο άλλο. Και εγώ. Κυρία Κάλλα, κυρία Κάπελ και μετά εγώ. Σα ευχαριστώ, γιατί είναι καλό να έχουμε και συμμετοχή από κυρίε. Ευχαριστώ. Με απασχολεί αυτό που είπατε για την αγορά και τις συστάσεις για να διευκολύνουμε την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στη λιανική πώληση. Με απασχολεί αν οι καταναλωτές θα έχουν τη σωστή πληροφόρηση. Αν γνωρίζουν τι προσφέρεται στην αγορά. Τι γνώμη έχετε για τα κομβικά σημεία δεδομένων που πρέπει να έχουν πάντοτε όλα τα TSO που επιτρέπουν στους καταναλωτές να γνωρίζουν πώς μπορεί να να κάνουν μετατόπιση από το ένα σύστημα στο άλλο. Οι διαχειριστές λοιπόν συστημάτων διανομής υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστούμε για Κάπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Λόρδε Μόκ και κύριο Ποτότσνικ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση αυτή. Σίγουρα έχετε επιλέξει την σωστή προσέγγιση να έχετε στο επικεντρό σας τον καταναλωτή. επικεντρώνεστε στους ιδιαίτερα ευάλωτους καταναρωτές ε, στην εκθεσή σας και είναι σημαντικό το μήνυμα που στέλνετε έτσι. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να τονίσετε περισσότερο τις δυνατότητες επιλογής που υπάρχουν. Ε, είπατε ότι αυτός είναι σημαντικός παράγοντας ε, για την διαμόρφωση των τιμών γιανικής. Κάτι άλλο που λείπει από την έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι οι φόροι και τα τέλη που επηρεάζουν την τιμή ενέργειας στα διάφορα κράτη-μέλη. Στην Αυστρία το ποσοστό των ε, τελών αυτών ανέρχεται σε 50% και είναι μεγάλο εμπόδιο για τον καταναλωτή. Ιδιαίτερα θα με ενδιέφερε, πέρα από την έκθεση αυτή για το 2014, θα ήταν ε, και η έκθεσή σας της 23 Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς ε, για την Αυστρία. Μη δεσμευτική σύστασή σας ε, ήταν ο διαχωρισμός κάτι όμως το οποίο θα προκαλούσε ε, κόστος ετήσιο 300, εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ζώνη όμως ε, για μας ε, είναι μια από τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ενέργειας. Αποτελεί υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας και ε, εφαρμόζεται εκεί και η αποθήκευση ενέργειας, κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε σήμερα. Στο γερμανικό δίκτυο, εάν ε, αυξήσουμε την ε, πίεση, δεν πρόκειται να βοηθήσουμε την κατάσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν εφαρμογή σωστών μέτρων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς ε, τη γνωμοδότησή σας της 23ης ε, ε, Σεπτεμβρίου. Θα εκπονήσετε μελέτη αντικτύπου και δεν πιστεύετε κι εσείς ότι αυτή η ζώνη αποτελεί μια από τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρτέλ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ μια ερώτηση για να με βεβαιώσω ότι καλά κατάλαβα. Ίσως παρανόησα, αλλά νομίζω είπατε ότι πρέπει η πώληση χομπρικής να πρέπει να αφήσει τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις για να υπάρξουν και πληστηριασμοί. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά, ίσως παρανόησα, αλλά δεν μπορούμε απλώς να ακολουθούμε την πολιτική του χαμηλότερου κόστου, τη τιμή μόνο. Η πολιτική των πληστηριασμών θα μπλοκάρει τις επενδύσεις. Θα είναι τροχοπέδι. Χρειάζονται έναν ορατό ορίζοντα οι επενδυτές και σήμερα η λύση αυτή δεν είναι και ιδιαίτερα διαδεδομένη. Παρανόησα λοιπόν ή αυτό είπατε. Αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα. Ευχαριστώ πολύ να προσθέσω κι εγώ κάτι. Σε όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ίσως κάτι γενικότερο. Διότι ήταν πολύ σωστή η αρχική σας δήλωση. Το πλέον σημαντικό για μας είναι οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές βρισκόνται στο επίκεντρο της δράσης μας. Τέλεια, πολύ ωραία. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, της οικονομίας μας και των επιμέρους καταναλωτών, των ε, εξτομικευμένων, των πολιτών δηλαδή. Όμως, χωρίς το τομέα της ενέργειας, πώς θα διοργανώσουμε την ενέργεια και θα υπερασπιστούμε τους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε τον κλάδο της ενέργειας. Άρα χρειαζόμαστε εταιρείε ενέργειας. Οπότε βεβαίως τελικώς απευθυνόμαστε στους καταναλωτές, αλλά μέσω των εταιρείων ενέργειας και στις δύο περιπτώσεις, και του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να συμβεί το εξή. Εάν συγκρίνουμε τι γίνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, στον τομέα του αερίου, οι τιμές μας, το κόστος, στην πώληση της χοντρικής και της λιανικής, είναι τουλάχιστον διπλάσιες τριπλάσιες από τις αμερικανικές. Θα παραδειγματιστούμε θα μας διευκολύνουν οι αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όμως είναι πολύ σημαντική η αγορά αυτή για την, ανταγωνιστικότητά μας. Για την ανταγωνιστικότητά μας. Πώς θα το προλάβουμε αυτό στον τομέα του αερίου ιδίω. Και μετά νομίζω ότι οι εταιρείε αερίου είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις Αμερικανικές στην Ευρώπη διότι θα πεθάνουν χωρίς επενδύσεις. Έχουν χαμηλές τιμές στις ε, σχεδόν ψυχοραγούν γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις. Τις επισκέφθηκα πρόσφατα τις ΗΠΑ, πριν από 15 μέρες. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η κατάσταση είναι κάπω κάπως διαφορετική. Στην αγορά λιανικής έχουμε λίγο πολύ παρόμοιες τιμές. Στην πώληση την χοντρική όμως, στη λιανική είναι πολύ ψηλότερες η κυρία Κάπελ είπε ότι όλες οι τιμές, έμεσο και άμεσο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλό. Και αυτό επιβαρύνει τον εθνικό προπολογισμό. Ιδίως το έμεσο κόστος. Να περιμένουμε από τους εθνικούς προπολογισμούς επενδύσεις, σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Διότι θέλουμε τον τομέα μας της ενέργειας. Ο συνάδελφος Μαρτά είπε ακριβώς το ίδιο. Πώς θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις στο τομέα της ενέργειας. Το υψηλό μέσο κόστος μάλλον θα καλύπτει τον εθνικό προπολογισμό. Πώς υπάρχει λοιπόν πώς μπορούμε να βρούμε δυνατότητα να στηρίξουμε τον τομέα της ενέργειας. Να φροντίζουμε με τους καταναλωτές ναι, αλλά με έναν ισχυρό τομέα ενέργεια και ισχυρέ εταιρείε ενέργεια. Σας ευχαριστώ όλους για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να πω κάποια πράγματα. Οι κρατικές ενισχύσεις νομίζω επίσης ε, θα αποτελέσουν ε, θέμα συζήτησης, αλλά σε επικεντρωθώ πρώτα στα πιο τεχνικά θέματα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να, καλε... να επιλέξουν αυτό που τους συμφέρει καλύτερα. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές. Καταρχάς, οι πληροφορίες σχετικά με τη δική τους ε, καταναλωτική συμπεριφορά και σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν τα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τον καταναλωτή να διατίθενται στον ίδιο τον καταναλωτή ή και σε άλλου εφόσον το επιλέξει ο καταναλωτή στον οποίο αφορούν τα δεδομένα. Η άλλη σημαντική πληροφορία είναι το τι υπάρχει στην αγορά. Και υπάρχουν κάποια εργαλεία σύγκρισης των τιμών κρατικών φορέων, ενώσεων καταναλωτών ε, και ιδιωτικών εταιριών. Και θα πρέπει να παρέχουν τα εργαλεία αυτά όχι μόνο τις σωστές πληροφορίες, κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά και συγκρίσιμες πληροφορίες. Ανέφερα, για παράδειγμα, τις μεγαλύτερες επιλογές που έχουν οι καταναλωτές, για παράδειγμα όσον αφορά το φυσικό αέριο, Υπάρχουν ε, πολύ περισσότερες προσφορές με πτυχή ε, βιωσιμότητας. Πώς μπορούν λοιπόν να συγκρίνουν οι καταναλωτές αυτές τις πληροφορίες. Κύριε Μάρτα, η έκθεση αυτή ασχολείται κυρίως με τις τάσεις βλέπουμε να υπάρχει μία τάση προς τιμολόγηση κόμβου και συμβάσεων μακράς διαρκείας. Αυτό δεν είναι κακό. Χρειαζόμαστε ενεργειακό τομέα πιο ευέλικτο και μια από τις προκλήσεις για το μέλλον είναι η ευελιξία. Χρειαζόμαστε ευελιξία και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο σύστημα. Και η ευελιξία έχει να κάνει περισσότερο με βραχυπρόθεσμες αγορές ε, παρά με συμβάσεις μακράς διαρκείας. Νομίζω λοιπόν ότι η τάση που βλέπουμε είναι μάλλον καλή. Άλλωστε συνήθως οι χρηματοπιστωτικές αγορές χειρίζονται τον κίνδυνο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό σημείο. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά και τι γίνεται με τις διαφορετικές ζώνες τιμών εάν το δυναμικό δεν μπορεί να στηρίξει μία ενιαία τιμή για όλους. Άκουσα διάφορες αντιδράσεις στη γνωμοδότησή μας. Σε μερικοί μου είπαν ότι δεν στηρίζεται την ενιαία αγορά. Βλέπουμε ότι αρκετές αγορές που λειτουργούν καλά εδώ και πολλά χρόνια έχουν διάφορες ε, ζώνες τιμολόγησης. Η Νορβηγία, η Ιταλία, πιο πρόσφατα η Σουηδία. Το θέμα είναι πώς οργανώνεται η αγορά. Εντός μιας ζώνης τιμολόγησης θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Αν είναι υπερβολικά μεγάλες οι ζώνες τιμολόγησης και αν δεν καλύπτονται από επαρκή υποδομή, τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε στρέβλωση της αγοράς. σε αθέμητα πλεονεκτήματα για κάποια είδη εμπορίου, ενώ θα, δεν θα πρέπει να έχουμε διακρίσεις. Εάν λοιπόν η υποδομή δεν είναι επαρκής ώστε να στηρίξει οι διάφορες, τιμές, οι ζώνες τιμολόγησης να, να θεωρηθούν μια ενιαία ζώνη, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Αναφερθήκατε λοιπόν ε, στην συνοριακή ζώνη Γερμανίας-Αυστρίας. Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής υποδομή για να ε, υπάρξει ενιαία ζώνη τιμολόγησης. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ κάτι για το άλλο σκέλος της ερώτησης, για, τους, για τις τιμές και τους δεσμούς για τα τέλη μάλλον. Ε, το καθαρό κόστος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της τιμής. Αν και είναι το μικρότερο, λιγότερο από το μισό του συνολικού κόστους τώρα η ηλεκτρική ενέργεια και επιδοτήσεις για τις ανανόμισιμες πηγές, οι φόροι, τα ποσοστά ΦΠΑ και το κόστος του δικτύου είναι το μεγαλύτερο μέρος της τιμής. Ανταγωνισμός λοιπόν για την ηλεκτρική ενέργεια ή για το αέριο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διότι για τις ανανεώσιμε πηγές έχουμε το ΦΠΑ και ε, την τιμή του δικτύου. Για το αέριο έχουμε γύρω στο 50% και για τον ηλεκτρισμό 40%. Οπότε είναι μεγάλο το ποσό. Συνέπεια είναι ότι ο ανταγωνισμό συμπιέζεται σε ένα πολύ στενό πεδίο περιορισμένο πεδίο. Νομίζω ότι το δικό σας σώμα ναι, υπάρχουν ανοιχτέ προκλήσεις αλλά νομίζω ότι πραγματικά το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει εάν πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις επιδοτήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και να έρθω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης του Πρόεδρου. Εάν τα επίπεδα φορολόγησης όπως ορίζονται από τις επιμέρους χώρες, χώρες είναι τα σωστά. Το μέσο όρο που έχουμε εντοπίσει είναι 15%. Με το ΦΠΑ όμως ε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε καμία αντίρρηση. Το να αυτά τα, τα τμήματα θα μειωθούν είναι κάτι που το αποφασίζουν οι εθνικές κυβερνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ τι κρατικέ βοήθειες. Και έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο σκέλος. Εάν θα μπορούσαν οι εταιρείε ενέργειας να επιδοτούνται κατά κάποιο τρόπο από τα κράτη-μέλη ως προς τις επενδύσεις τους κυρίως. Διότι τα πορεία οικονομικών από την μια παίρνουν ε, πολλά κονδύλια στα χέρια του. Κάποια από αυτά θα έπρεπε να τα προωθούν στι ε, εταιρείε ενέργεια για, την... Ε, για τι επενδύσει. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Και το δεύτερο δεν νομίζω ότι θα ήταν αναγκαίο. Νομίζω ότι αυτό που είναι αναγκαίο είναι αυτό που έχουμε σε ορισμένε χώρε και συμβαίνει ήδη. Μια ένα τέτοιο αυστηρό νομοθετικό καθεστώς που εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν. Το λέω εδώ και χρόνια. Ίσως να μην είχα πάντοτε δίκιο, αλλά αυτή τη φορά νομίζω πως ναι. Υπάρχουν κεφάλαια διαθέσιμα για να επενδυθούν είναι διαφορετικό να υπάρχουν κακέ επενδύσει από τον κρατικό φορέα γιατί εξυπηρετούνται διαφορετικοί σκοποί. Διαφέρει από τους επενδυ... να βλέπουν οι επενδυτέ να υπάρχει ένα σταθερό σύστημα παρά διαρκεί μετακινήσει, μετατροπέ, αυξημένοι φόροι κτλ. Αυτό το κλίμα είναι που εμπνέει του επενδυτέ. Τώρα, οι υποδομέ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ε, αυτέ δεν παροτρύνουν αναγκαστικά του επενδυτέ. Και τελευταίο σημείο, θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για το θέμα αυτό. Είναι ακριβώ αλήθεια αυτό που λέτε, Πρόεδρε, ότι το αέριο και το κλάδο του αερίου έχει πληγεί πάρα πολύ από τι χαμηλότερε τιμέ στι ΗΠΑ. Η διαφορά είναι το σχιστολιθικό αέριο από την Ευρώπη. Οι Αμερικανοί εξάγουν το σχιστολιθικό σε μεγάλες ποσότητες και αυτό επηρεάζει το κόστος εδώ. γιατί δεν είναι και απλή η διαδικασία του στο αέριου αέριο της Αμερικής να φτάσει ως εγώ, νομίζω. Ε, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες επωφελήθηκαν από το σχιστολιθικό αέριο για πολύ καιρό, όπως έγινε με το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 60 που είχε αποφεληθεί τότε από την αγορά αερίου. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα υπάρξει λιγότερη, λιγότερο ενδιαφέρον να εξαχθεί προς εδώ το αέριο αυτό, οπότε ίσω και περισσότερα προβλήματα για τον κλάδο του αερίου στι ΗΠΑ. Η σύντομη απάντηση είναι ότι πάρα πολλά από την σκοπιά της ενέργειας ταπανώνται σε στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά αυτά πρέπει να τα αποφασίσουν οι εθνικές κυβερνήσει, το Κοινοβούλιο και άλλοι. Οι επιδοτήσει είναι πάντοτε ένα κίνδυνο για οποιοδήποτε σύστημα και το βλέπουμε διαρκώ αυτό να συμβαίνει, αλλά πρέπει κανείς να εξορροπήσει τα ωφέλη και τι ζημιές. Ε, πρόεδρε, πρέπει κανεί να διαλέξει το σωστό σημείο ισορροπία ή την ανάγκη να υπάρχουν νέε πηγέ ανανεώσιμη ενέργειας, αλλά το σχιστολήθικο ε, είναι ένα αμερικανικό φαινόμενο, μπορεί να παραμείνει τέτοιο. Το αν θα αλλάξει τη ζωή των εταιριών ή όχι, θα φανεί. Εγώ αμφιβάλλω. Ελπίζω οι τεχνικοί που τις Επιτροπής που μας ε, βλέπουν να μην έχουν φρίξει με τις απαντήσεις μου. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα ξανασυναντηθούμε έτσι και αλλιώς και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τους καταναλωτές στο επίκεντρο της προσοχής μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείε ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αρκετά δυνατές για να διοργανώσουμε σωστά την αγορά μας και να ε, παρέχουμε ασφαλή ενέργεια στους καταναλωτές μας. Να προσθέσω συνάδελφοι, πάρα πολύ σημαντικό, ότι ότι η δική μας συζήτηση εξυπηρετεί πολύ και την Άσερ, διότι μετά τη συζήτησή μας και την ψήφο στην Ολομέλεια, 15 νέες θέσεις εργασίας εμφανίστηκαν στην Άσερ, χάρη στη δική μας την παρέμβαση. Φανταστικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι ήταν απολύτω αναγκαίο, εάν θέλετε να είστε κι εσεί επιτυχημένοι για την αγορά ενεργειά μα, να μπορείτε να δουλέψετε σωστά. Ευχαριστούμε λοιπόν, ευχαριστούμε για όλε σα τι ε, ε δραστηριότητε. Ευχαριστώ συνάδελφοι, θα συναντηθούμε αύριο στι 10. 10. Ευχαριστώ.